So, ladies and gentlemen, good morning. Welcome to all of you. First of all... Καλημέρα, καλώς ορίσατε όλοι κυρίες και κύριοι. Καλώς, ε, καλώς ορίσατε υποψήφια επιτροπή κυρία Κάντρι Σίμψον. Το χαρτοφυλάκιο σας προτάθηκε όπως προτάθηκε από την ε, νέα πρόεδρο την κυρία Λάιεν, είναι το χαρτοφυλάκιο ενέργειας. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ στην αίθουσα τα μέλη της Επιτροπής ΙΤΡΕ, ΕΜΒΗ η οποία επίσης ε, παρίσταται σε αυτή την ακρόαση. Η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά με web streaming. Καλωσορίζουμε λοιπόν και όσους μας ε, παρακολουθούν μέσω διαδικτύου. Η Επιτροπή Ήτρε είναι αρμόδια για την ενεργειακή πολιτική της Ένωσης. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ενέργεια διαδραματίζει ένα ρόλο κλειδί στην κοινωνία μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει πλήρω και τι πέντε διαστάσει τη Ενεργειακή Ένωση. Ενεργειακή ασφάλεια, εσωτερική αγορά ενέργεια, ενεργειακή απόδοση, απαλλαγή από ανθρακούχε εκπομπέ, έρευνα, κοινοτομία και ανταγωνιστικότητα. Η ενέργεια έχει να παίξει σημαντικό ρόλο ε, στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου, του European Green Deal, που θα παρουσιαστεί εντός των πρώτων 100 ημερών της Νέας Επιτροπής και θα βρίσκεται στο επίκεντρο της θητείας της. Να σας υπενθυμίσω πώς θα διεξαχθεί η σημερινή ακρόαση. Σύμφωνα με τις κατευθύντηρες γραμμές για την έγκριση της Επιτροπής, το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους υποψήφους επιτρόπους βάσει των γενικών ικανοτήτων τους, της ευρωπαϊκής τους δέσμευσης και της προσωπικής τους ανεξαρτησίας. Επίσης αξιολογεί τις γνώσεις τους όσον αφορά το σχετικό τους χαρτοφυλάκιο και τις ε, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Οι εργασίε μα σήμερα οργανώνονται ως εξής. Πρώτα απ' όλα υποψήφια θα πραγματοποιήσει σε 15 λεπτά μία παρουσίαση. Θα έχουμε ένα γύρο ερωτήσεων από, πρώτα από τις πολιτικές ομάδες, μετά από τα υπόλοιπα μέλη, σύμφωνα με το σύστημα DEONT. Κάθε ερώτηση μπορεί να διαρκεί 5 λεπτά, ε, ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση, ε, ένα λεπτό για δευτερολογία και ένα λεπτό για τη δεύτερη απάντηση. Η δεύτερη ερώτηση πρέπει να αναφέρεται στο ίδιο θέμα με την πρώτη. Θα είμαι αυστηρή με τους χρόνους, οπότε παρακαλώ προσέξτε ε, τις ερωτήσεις σας ε, και τις απαντήσεις σας, ώστε να τηρούμε τους χρόνους. Τους χρόνους τους βλέπουμε στην οθόνη, μπορείτε να τους ε, δείτε να πάσα στιγμή. Κυρία Καντρί Σίμψον, ε, θέλω να σας καλωσορίσω. Έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Σα ευχαριστώ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε Βαλεάν ε, και Ευρωβουλευτές τη ε, της Επιτροπής Βιομηχανίας Περιβάλλοντος, σας ευχαριστώ. Είμαι, χαίρομαι που είμαι σήμερα εδώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά για μένα είναι σίγουρα η πιο σημαντική. Ε, με τιμά η απόφαση της υποψηφίας Προέδρου Ούρσουλα Φαντελάιεν να επιλέξει εμένα ως υποψήφια επίτροπο αρμόδια ε, για την ενέργεια. Και είναι σήμερα η τιμή μου να σας παρουσιάσω ποια είναι τα σχέδιά μας για την ενέργεια. Οι χιλιάδες άνθρωποι που κατεβαίνουν στους δρόμους ε, μας θυμίζουν ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο επίγον από ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι υπαριθμόν ένα έρημνα και ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό και η υποψήφια Πρόεδρος έχει εντοπίσει την ε, ε, ε, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως πρωταρχικό στόχο. Η ενεργειακή πολιτική θα είναι ύψη της σημασίας ώστε να αποδώσει αυτή η προτεραιότητα. Ήμουν, έχω διατελέσει υπουργό Οικονομίας και Υποδομών, υπεύθυνη επίσης για την ενέργεια στη χώρα μου και ξέρω πόσο μεγάλη πρόκληση είναι τα θέματα αυτά πόσο σημαντικό είναι το έργο που μας αναμένει και πόσο τεράστια η ευθύνη τα τελευταία πέντε χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει τεράστια άλματα προς την Ενεργειακή Ένωση στις πέντε της διαστάσεις. Όλα τα μέτρα του δέσμης για την καθαρή ενέργεια που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο είναι μια σπουδαία, ένα σπουδαίο κληροδότημα επί το οποίο θα μπορούμε να βασιστούμε. Θέλω γι' αυτό να ευχαριστήσω τον αρμόδιο επίτροπο Αρέας Κανιέτε και τον αντιπρόεδρο Σεφτσοβίτς που μας ε, οδήγησαν σε αυτό το σημείο στο οποίο ε, βρισκόμαστε σήμερα, αλλά να ευχαριστήσω και τις επιτροπές σας που συνέβαλαν ώστε να σημειωθεί αυτή η πρόοδος. Χάρη σε εσά το Ευρωκοινοβούλιο ε, αυξήθηκε το επίπεδο φιλοδοξίας του αρχικού ε, πακέτου για την καθαρή ενέργεια και επίσης συμβάλλατε στο να εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία. Αυτό δείχνει την αξία της ενότητας. Όταν είναι, είμαστε ενωμένοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικές αλλαγές. Αλλά εδώ τώρα ε, δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε στις ε, δάφνες μας. Το να επιτύχουμε τους στόχους για το 2050 είναι ο μόνος τρόπος να περιορίσουμε στον 1,5 βαθμό την αύξηση της δημοκρασίας και να προλάβουμε την περιβαλλοντική κρίση. Και γι' αυτό και η υποψήφια πρόεδρος ε, υποσχέθηκε να ε, καταστήσει την Ευρώπη καθαρή ήπειρο μέχρι το 2050 και να προτείνει μια πράσινη ε, συμφωνία, Green Deal, για ενώπιον του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Εγώ θα ήθελα να σας εκθέσω πώς σκοπεύω να προχωρήσω στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική ως Επίτροπος. Ε, συμφωνώ στον, φυσικά στον στόχο του να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ήπειρος ουδέτερη προς το κλίμα μέχρι το 2050 και να περιοριστούν κατά 70% οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030. Ε, η Εστονία αυτή τη στιγμή ε, θα ξεπεράσει μάλλον τους προβλεπόμενους στόχους. 42% το 2030 θα φτάσουμε και έχω μάθει ότι η διαδικασία μετάβασης μπορεί να λειτουργήσει σωστά όταν γίνονται σαφείς επιλογές. Πρώτα απ' όλα αυτό που χρειάζονται οι φορείς στην ενέργεια από, τον, από τους ρυθμιστές είναι η βεβαιότητα και η προβλεψιμότητα έτσι ώστε να μπορούν να προγραμματίσουν σε πρώιμα στάδια. Γι' αυτό και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ε, ε, μια πράσινη συμφωνία στα πρώτα, στις πρώτες 100 μέρες θητείας. Να Νέα νομοθεσία που θα θεσπίσει την ουδετερότητα στόχο για το 2050 δεχόμαστε και αυτή την ε, κατεύθυνση και θα πρέπει να βασιστούμε στην επιτυχία της Ενεργειακής Ένωσης. Η Εστονία έχει τη, τη φήμη ότι είναι ε, χώρα που κοιτά συνέχεια προς το μέλλον. Εγώ δεσμεύομαι να εργαστώ σκληρά για την εφαρμογή του πακέτου για την καθαρή ενέργεια. Θα εξασφαλίσω πως τα κράτη-μέλη θα υιοθετήσουν φιλόδοξα εθνικά σχέδια μέχρι το τέλη του ε, Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειμμα αφιλοδοξίας θα κάνω κάθε προσπάθεια να οθήσω τα κάτι μέλη προς τη σωστή κατεύθυνση και θα τους παροτρύνω για να, όλους για να επιτύχουμε τους στόχους. Πρέπει να προσαρμόσουμε το δυναμικό αυτό της, ε, του καθαρού πακέτου για όλους τους ε, Ευρωπαίους. Ε, πρέπει να υιοθετηθούν ακόμα πάνω από 100 εφαρμοστικές πράξεις. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Εφαρμόζοντας τις ίδιε χιούσες νομοθεσίες μπορούμε να περιορίσουμε κατά 40% τι εκπομπές μέχρι το 2030. Η υποψήφια πρόεδρος είπε ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι όταν μιλάμε για τους στόχους του 2030. Δεσμεύτηκε για περιορισμό των εκπομπών τουλάχιστον του τάξη του 50% μέχρι το 2030 θα ξεκινήσουμε μια αξιολόγηση για το πώς ε, μπορεί να αποδώσει ε, και να επιτύχει πιο φιλόδοξους στόχους η νομοθεσία περί ενέργειας. Και με βάση αυτή την αξιολόγηση θα ξεκινήσουμε νέες ε, νομοθεσίες. Αναθεώρηση της οδηγίας περί φορολογίας της ενέργειας που προτάθηκε από τον Παόλο Τζεντιλόνι. Θέλουμε επίσης περαιτέρω να αναπτύξουμε και να ολοκληρώσουμε μια ορθά λειτουργούσα ενιαία αγορά. Μια τέτοια εσωτερική αγορά επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα και επιτρέπει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, πιο γρήγορα. Εγώ ως υπουργό έχω εργαστεί για το δίκτυο των βαλτικών χωρών και τη σύνδεση αυτών με την, με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είδαμε πως ένας καλός συντονισμός είναι προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, την ασφάλεια στην ενέργεια και την επάρκεια ανεφοδιασμού και ελπίζω πως αυτά όλα θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος αυτής της αιτίας. Δυστυχώς οι ολοκληρωμένες αγορές δεν είναι ο κανόνας ολόκληρη την Ευρώπη. Στον τομέα της, του ηλεκτρισμού χρειάζεται ένα σύστημα ε, παραγωγής που θα βασίζεται στις ανανεώσιμες, στην αυξημένη ε, διασύνδεση και ε, της, ε, τη δυνατότητα σώρευσης και αποθήκευσης της ενέργειας. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε πως οι στόχοι διασυνδεσιμότητα θα επιτευχθούν και το 70% των δυνατοτήτων διασύνδεσης θα ε, επιτευχθεί ε, σύντομα. Εγώ δεσμεύομαι να ενισχύσω την διαπεριφερειακή συνεργασία και ε, προωθώντα την εργασία των τεσσάρων intergroup για αυτή τη δουλειά, για αυτούς τους στόχους. Θέλω να επικεντρωθώ και στο φυσικό αέριο για να βελτιωθεί το δίκτυο ε, και να είναι έτοιμο για το μέλλον και οι υποδομές για την ε, απομάκρυση από το διοξίδιο του άνθρακα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε υδρογόνο και ανανεώσιμες. Ε, θα πρέπει ε, να είναι και προς όφελος των τελικών καταναλωτών οι δυνατότητες που έχουμε με το υγροποιημένο φυσικό ε, αέριο. Έχουμε επιτυχή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να συνεχιστεί. Η ολοκλήρωση της αγοράς είναι επίσης μια πρόκληση για τις υποδομές. Χρειάζονται 250 δις περίπου μέχρι το 2030 για να κλείσουν οι βρόχοι ε, και ε, να υπάρξει αλυσίδα του εφοδιασμού. Ε, θα πρέπει να βασιζόμαστε στην καλύτερη αποθήκευση ενέργειας, στις ανανεώσιμες και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες των δικτύων. Για να γίνει αυτό, μέχρι το 2020 θα έχω ολοκληρώσει την αξιολόγηση των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας. Είναι τεράστια επίσης πρόκληση η χρηματοδότηση. Θα πρέπει να βρούμε και να μοχλεύσουμε και ιδιωτικούς πόρους. Ε, με το επόμενο ε, στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα έχουμε 122,2 δις. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Θα πρέπει να βελτιωθεί η ε, ενεργειακή απόδοση των κτηρίων για να αλλάξει πραγματικά ε, η νοοτροπία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια, αλλά μπορούμε να βρούμε λύσεις για τη χρηματοδότηση. Με καλά παραδείγματα που υπάρχουν σε πολλά κράτη-μέλη στην κοινωνική στέγη και σε τοπικό επίπεδο. Επίσης μπορούμε να γίνουμε κλιματικά ουδέτεροι διατηρώντα την ανταγωνιστικότητά μα ταυτόχρονα και της βιομηχανίας. Υπάρχουν ποιοτικέ θέσει εργασίας στις ε, καθαρές τεχνολογίες εάν η Ευρώπη είναι ηγέτης. Ε, υπάρχει τρόπο για ευφύ καινοτομία ε, στον ηλεκτρισμό, στην θέρμανση, στις μεταφορέ κτλ. Και τέλος, θα ε, προσέξω και τις τιμές της ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή, είτε είναι νοικοκυριά είτε είναι βιομηχανίες, ε, για να ε, προχωρήσουμε στην κλιματική μετάβαση. Εγώ είμαι φιλελεύθερη. Ανέκαθεν επίστευα στις προσωπικές ελευθερίες, χωρίς να λησμονώ τη δικαιοσύνη. Η κλιματική μετάβαση θα επηρεάσει πολλούς και βαθιά και κάποιους περισσότερα από κάποιους άλλους. Μπορώ να σας παραθέσω στατιστικές, αλλά αυτά δεν είναι μόνο αριθμοί. Πρόκειται για ανθρώπους και έχουν και ζωές και έχουν και ιστορίες οι άνθρωποι αυτοί. Ολόκληρες οικογένειες, ε, χωριά, από τη Γαλλικία μέχρι τη Σιλεσία ε, θα γνωρίσουν μεγάλες αλλαγές. Το καταλαβαίνω αυτό από πρώτο χέρι, γιατί είμαι από την Εστονία. όπου χρησιμοποιείται ευρέως ακόμα ο ε, άνθρακας. υπάρχει μια πρόβλεψη για να υποστηριχθούν οι περιφέρειες που εξαρτώνται από τον άνθρακα και τα νησιά. Και μια, είναι μια ιδέα αυτή που ξεκίνησε από το Κοινοβούλιο. Και είμαι βεβαία ότι το θυμάται πολύ καλά αυτό ο καθηγητής Μπούζεκ. Το ταμείο αυτό θα βοηθήσει τις περιφέρειες να αναπτυχθούν, να αναπτύξουν και να χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένα έργα που θα μετασχηματίσουν τις οικονομίες τους και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Υπάρχει μια τέτοια πρωτοβουλία και θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε για να γίνει επιτυχία αυτό το ταμείο. Επίσης θα πρέπει να εντείνουμε τον αγώνα μας ε, για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. 15 εκατομμύρια ε, πολίτες, το 8% του πληθυσμού, ε, δεν μπορούν, ε, μάλλον 50 εκατομμύρια, δεν μπορούν να ε, ζεσταθούν και να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Υπάρχει μεγάλο θέμα με την ενεργειακή φτώχεια. Θέλω να συνεργαστώ καλύτερα με τα κράτη-μέλη και τους Δήμους. Η Τερέζα Κρίφιν πέρσι κατέθεσε μια έκθεση που έβαλε τα θεμέλια για την υπόθεση αυτή. δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι θα είμαστε στην Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050 χωρίς να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες. Ε, είμαστε ε, ένας γίγαντας ε, στην έρευνα, δεύτερη μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, με μεγάλη έρευνα, με πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αλλά οι επενδύσεις δεν ε, ακολουθούν. Θα συνεργαστώ με τη συνάδελφο Μαρία Γκάμπριελ για να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη προς την κατεύθυνση αυτή. Το στρατηγικό τεχνολογικό πρόγραμμα έχει δυναμικό και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε πλήρως. Σκέφτομαι να ε, καταρτήσω ένα θεματολόγιο για τη μεγαλύτερη ψηφιοποίηση ε, της ενεργειακής αγοράς, καλύπτοντας την ψηφιακή αγορά, την καθαρή, ε, τα εφή δίκτυα, την πρόσβαση και τη διαλειτουργικότητα. Αλλά επίσης την κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη η ε, Ευρώπη θα πρέπει να πιέσει και άλλους ε, ρηπαντές, ε, χώρες που εκπέμπουν πολλούς ρήπους, να ακολουθήσουν τη Συμφωνία του Παρισιού. Και επίσης φυσικά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τον ανεφοδιασμό μας. Έχει έρθει η ώρα να ενισχύσουμε και το κοινό μας νόμισμα και τα ενεργειακά συμβόλαια να γίνονται περισσότερο σε ευρώ πλέον. Στην Ουκρανία έχουμε διμερή ε, ε, συμφωνία και θα πρέπει να καταλήξουμε μέχρι τα τέλη του έτους. Για πολλά χρόνια διετέλεσα μέλος του Εστονικού Κοινοβουλίου Γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι προτίθεμαι να συνεργαστώ πάρα πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εξηγώ κάθε φορά τι κάνουμε ε, όταν έχουμε νέες εξελίξεις. Θα είμαι στη διάθεσή σας. Μεγάλωσα στην Εστονία. Όταν η Ευρώπη ήταν όνειρο, ιδεώδες, ελπίδα για αλλαγή και ελευθερία. Εγώ πιστεύω στην Ευρώπη και θέλω να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου σε μια Ευρώπη που να φιλοδοξεί για περισσότερα με αποφασιστικότητα αλλά και ταπεινότητα ταυτόχρονα. Ε, υποστηρίζω στη δική σας, μάλλον προσβλέπω στη δική σας υποστήριξη και ε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την Ευρώπη στα ενεργειακά και στα κλιματικά ζητήματα. Uh, λοιπόν, και τώρα έχει έρθει η ώρα των ερωτήσεων από τα μέλη των επιτροπών μας, της Ήτρε και Ένβη. Θυμίζω ότι έχουμε ένα πεντάλεπτο ping-pong. Ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση, ένα για τη συμπληρωματική ερώτηση, ένα για τη συμπληρωματική απάντηση. Ο κύριος Μπούζεκ πρώτος ε, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την ομιλία σας, κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Την τελευταία πενταετία έχουμε επιτύξει πολλές προσπάθειες ε, ολοκλήρωσης της Ενεργειακής Ένωσης. Τώρα η πρώτη μας προτεραιότητα είναι χωρίς άλλη καθυστέρηση να υλοποιήσουμε ε, τα νομοθετικά, τα νομοθετήματα. Η ενεργειακή μετάβαση θα αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα Δίκαιοι θέλουμε να είναι μετάβαση, ε, είναι πολύ σημαντικό. Αναμένω να παίξετε σημαντικό ρόλο εδώ και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τις διάφορες επενδύσεις σε, ε, σε ενέργεια ε, χαμηλών εκπομπών, την τηλεθέρμανση, τις υποδομές από πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιωτικούς πόρους, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Πώς θα διασφαλίσετε ότι θα αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το φυσικό αέριο στην ενεργειακή μετάβαση. Ευχαριστώ κύριε Σίμψον. Ευχαριστώ κύριε Μπουζε για την ερώτησή σας. Πριν απαντήσω, επιτρέψτε μου να τονίσω για άλλη μια φορά πόσο σημαντική ήταν η Επιτροπή η και εσείς προσωπικά στις ε, διαπραγματεύσεις ε, που προηγήθηκαν για το πακέτο καθαρή ενέργεια. Δεν μπορώ παρά να επιβεβαιώσω λοιπόν ότι η δουλειά που έγινε αποτελεί ένα εξαιρετικό θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε. Ρωτήσατε για τη μελλοντική χρηματοδότηση. Πράγματι αληθεύει. Αν ε, Έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους. Το μεγαλύτερο εμπόδιο, ειδικότερα για τα έργα ενεργειακής απόδοσης, είναι η χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα, οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα περιλαμβάνουν ως βασική προτεραιότητα τις κλιματικές επενδύσεις. Έτσι αναμένουμε ότι θα υπάρχουν περισσότερα κονδύλια διαθέσιμα για έργα ενεργειακής ε, απόδοσης, για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για δίκτυα επίσης. Στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται ανάλυση των μελλοντικών ε, δανειοδοτικών ε, διαδικασιών και καλό είναι ότι θα υπάρξει αυτή η κλιματική τράπεζα που θα μας δώσει περισσότερα κονδύλια για επενδύσεις και σας υπόσχομαι ότι εγώ θα συνεργαστώ πολύ στενά με τον Επίτροπο Τζεντιλόνη και θα έχω ε, τακτικές επαφές με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ούτως ώστε τα νέα ε, κριτήρια δανειοδότησης να είναι σύμφωνα με τους κλιματικούς μας στόχους. Και τις Ευρωπαϊκές Αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπούζεκ. Ευχαριστώ αξιότιμη κυρία. Ήθελα να πω η τηλεθέρμανση είναι πολύ σημαντική από αυτή την άποψη και η ε, αυτόνομη θέρμανση. Λοιπόν, τώρα η ερώτησή μου είναι για τον τομέα του φυσικού αερίου. Διότι έχουμε την αναθεώρηση ε, ε, τη οδηγία, την δηλώσαμε την αναθεώρηση τη οδηγία για το φυσικό αέριο στην προηγούμενη θητεία. Και τώρα θα υλοποιηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία στην ευρωπαϊκή επικράτεια για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα του φυσικού αερίου. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια νέα όθηση σε αυτό το μέτωπο. Και ήθελα να σα ρωτήσω, είστε έτοιμοι για την πλήρη υλοποίηση της αναθεώρησης της οδηγίας για το φυσικό αέριο παρά των διαμαρτυριών της Ρωσίας, γιατί ξέρουμε από πού προέρχονται οι διαμαρτυρίες. Διότι θα βοηθούσε πάρα πολύ και την τηλεθέρμανση και την ε, αυτόνομη θέρμανση σε τουλάχιστον 15 κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κύριε Σίμψον. Ευχαριστώ κύριε Μπούζε και πολύ σωστά είπατε ότι το φυσικό αέριο είναι σημαντικό εργαλείο για την μεταβατική περίοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή για την τηλεθέρμανση. Και θα παραμείνει σημαντικό. Πρόκειται μάλλον για την πιο οικονομικά αποτελεσματική επιλογή αντικατάστασης ε, του κάρβουνου και των σχετικών εγκαταστάσεων. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μελλοντικέ ενεργειακές πηγές πρέπει να είναι διαφοροποιημένες. Οπότε όταν μιλάμε για φυσικό αέριο, στο άμεσο μέλλον δεν μιλάμε μόνο για φυσικό αέριο, αλλά και για βιολογικά αέρια και για υδρογόνο που μπορούν να μας βοηθήσουν να υπερβούμε ε, κάποια προβλήματα, ειδικότερα όσον αφορά τη θέρμανση, την ψήξη, ε, τη χρήση βιομηχανικής ενέργειας ή τις μεταφορές. Ε, ευχαριστώ. Thank you. Um, next speaker is Mr. ο κύριο Τζορίνιο, επόμενο από τη Σοσιαλιστή και Δημοκράτες για την Επιτροπή Βιομηχανίας. Καλημέρα σας κυρία υποψήφια επίτροπε. Αν θέλουμε να κάνουμε ψηφιακή την οικονομία μας, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να λαμβάνουμε υπόψη τις διάφορες πραγματικότητες. Δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε ε, απέναντι στις κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια ψηφιακή μετάβαση. Η δίκαιη μετάβαση ήταν και παραμένει προτεραιότητα των σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πείσαμε και την ε, κυρία Φόντερ Λάιεν, ε, το δήλωσε και η ίδια στην ομιλία της. Προβλέπεται και ένα ταμείο για την ε, δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και θα συνεργαστείτε και με την κυρία Φερέιρα, την ε, αρμόδια επίτροπο. Ω επίτροπος ενέργειας, λοιπόν, πώς προτίθεστε να βοηθήσετε για την ενεργειακή πολιτική, ακριβώς να βοηθήσετε την κυρία Φερέιρα στο έργο που θα έχει να επιτελέσει. Και δεύτερη ερώτηση. Το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση θα είναι και κοινωνικής πολιτικής για να βοηθάει εκείνους που θα πληγούν περισσότερο ή όχι μόνο αυτό θα προωθεί και την καινοτομία για να έχουμε μια δίκαιη, επαναλαμβάνω, ενεργειακή μετάβαση. Ευχαριστώ κύριε Ζωρίνιο για την ερώτηση. Το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση βεβαίως θα μου είναι πάρα πολύ προσφυλές γιατί είναι το εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εξασφαλίσουμε ε, τη μετάβασή μας προς την ουδετερότητα σε σχέση με τον άνθρακα και δεν θα πρέπει να μείνει πίσω ούτε μία χώρα ούτε μία περιφέρεια. Ως εργαλείο το βλέπω και το θεωρώ χρήσιμο για να φτάσουμε στο στόχο μας. Έτσι ώστε ε, οι περιοχές που εξαρτώνται από τον άνθρακα ή από άλλα ορυκτά καύσιμα, καθώς επίσης και μικρά νησιά που δεν έχουν καλές συνδέσεις με την ε, ενδοχώρα, με την υπηρετική χώρα, να μην ε, μείνουν πίσω. Αυτές οι περιφέρειες όμως δεν είναι ομοιογενείς. Έχουν μεγάλες διαφορές δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία λύση, κουστούμι για όλες τις περιφέρειες. Στρατηγικές θέλουμε για να δούμε πώς θα προετοιμαστούν καλύτερα για να καλύψουμε το στόχο μας. Δηλαδή θα είναι κάθε λύση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της εκάστοτε χώρας ή περιφέρειας. Αυτό λοιπόν το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση, ξέρω ότι θα το προτείνει η Επίτροπος Φερέιρα, αλλά δεν θα πρέπει να κινητοποιεί μόνο τις υπάρχουσες δυνατότητες. Χρειάζεται και υποστήριξη των κρατών μέλων και επιπλέον χρηματοδότηση. Το μεγαλύτερο ατού του ταμείου αυτού είναι ότι θα αρχίσει να λειτουργεί πριν τη φάση εκπνοής, αυτό το phasing out θα δώσει στις βάλλοντες αυτές περιφέρειες ένα σχέδιο για το μέλλον. Πριν χαθούν οι εξορεκτικές ε, δραστηριότητες και οι αντίστοιχες θέσει εργασίας. Για να ανοίξουν νέες ευκαιρίες για τις περιφέρειες αυτές. Ευχαριστώ. just an indication that you're... Ε, μάλιστα. Αυτό αυτό μας δείχνει ότι ασχολείστε τόσο πολύ με αυτά. Ε, ε περώτηση, κύριε Ζωρίνια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν υπάρχει αφιβολία ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις, ειδικά στις ε, περιφέρειες και στις κοινωνίες με πρότυπα παραγωγής ενέργειας τα οποία είναι πιο ρηπογόνα. Όμως δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρξει σύγκληση. Σύγκληση ε, που να έχει νόημα για όλους τους Ευρωπαίους να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην τεχνολογικό άλμα για ολόκληρη την Ευρώπη. Ξέρω πως είναι δύσκολο αυτή τη φάση να μιλάμε για νούμερα, απλά θέλω να ξέρω ποιο είναι το επίπεδο φιλοδοξίας σας. Αν συμφωνείτε με την αρχή ότι οι νέες πολιτικές ε, πρέπει να συνοδεύονται από νέα κονδύλια ε, και λαμβάνοντας υπόψη το Κοινοβούλιο στην πρόταση του επόμενου πολιετούς ε, χρηματοδοτικού πλαισίου προτείνει ε, μεγάλο κονδύλι Ξέρετε ότι γίνεται ένα κομμάτι από τις επενδύσεις ε, με βάση δάνεια, αλλά πιστεύετε πως αυτό το κονδύλι που προτείνει το Κοινοβούλιο είναι αρκετό, είναι μια καλή βάση. Ε, η κυρία Σίμψον, ευχαριστώ. Ναι. Πιστεύω πως αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι ένα συγκεκριμένο μέτρο για να βοηθηθούν εκείνες οι περιφέρειες οι οποίες θα επηρεαστούν περισσότερο λόγω της σταδιακής ε, ε, εξάλληψης της εξόριξης άνθρακας και των λοιπόν στερεών καυσίμων ορυκτών, με συγχωρείτε, καυσίμων. Υπάρχουν ε, διάφορα μέτρα που μπορούν να δώσουν πιο ανταγωνιστικές ε, ε, τιμές και αυτό είναι κομμάτι της διαδικασίας πάυσης χρήσης του άνθρακα για να μπορούμε να έχουμε ασφαλή σπόρους αλλά για τις περιφέρειες όπου οι, τοπικά παρα... Ε, τοπικές ανανεώσιμες δεν χρειάζεται να είναι τόσο πολύ δαπανηρές αλλά δεχόμενοι και ότι υπάρχουν διακοιμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, μπορούμε να προβλέψουμε ε, επενδύσεις που θα επιτρέψουν στις τοπικές ε, κοινότητες να φροντίσουν για την ε, παραγωγή ενέργειάς τους και για την επάρκεια σε ενέργεια, ώστε δηλαδή οι καταναλωτές να χρειάζεται να δαπανούν λιγότερη ενέργεια από ό,τι τώρα. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Πέτερσεν, ε, μέλος της ΙΤΡΕ από το Renew Europe. Ευχαριστώ, θα μιλήσω δανέζικα. Ε, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την... τις άριστες ε, και πλήρεις γραπτές απαντήσεις που λάβαμε στην Επιτροπή μας. Τις διαβάσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω μία ερώτηση για την βιώσιμη ενέργεια για να έχουμε κλιματική ουδετερότητα στην Ευρώπη μέχρι το 2050. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι αυτή τη στιγμή. Αλλιώς δεν θα επιτύχουμε τους ε, στόχους. Η τιμή της αιωλικής και της ηλιακής ενέργειας έχει πέσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, το οποίο σημαίνει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς επιδοτήσεις σε μεγάλο βαθμό. Ίσως αυτή να αποτελήσει μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις. Αν η εστίαση λοιπόν στις ανανόσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση. Έχουν... Η ολική ενέργεια της Ευρώπης είναι από τις καλύτερες του κόσμου. Μπορούμε να ανταγωνιστούμε την Μέση Ανατολή αν εστιαστούμε σε αυτήν. Αλλά θα χρειαστεί να αξιοποιήσουμε περισσότερο τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα, πέντε φορές περισσότερο από ό,τι αυτή τη στιγμή. Τι λέτε να γίνει με αυτό στη Βόρεια Θάλασσα ειδικότερα. Ευχαριστούμε κυρία Σίμψον. Ευχαριστώ κυρία Πέτρισεν για την ερώτησή σας. Συμφωνώ μαζί σας. Χρειαζόμαστε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περισσότερες δυνατότητες από αυτές. Και ξέρετε αυτές οι νέες εγκαταστάσεις πρέπει να την χάνουν και δημόσια αποδοχής, ε, τα υπεράκτια αιωλικά πάρκα τείνουν να είναι πιο αποδεκτά από τον κόσμο από ότι τα επίγεια. Ε, δεδομένου ιδιαίτερα ότι οι καλύτερες ε, τοποθεσίες έχουν ήδη καταληφθεί οι επίγειες τοποθεσίες. Θεωρούμε ότι θα χρειαστεί στενή συνεργασία μεταξύ των διαφορών κρατών μελών <laughs> για την κατασκευή των νέων υπεράκτιων εγκαταστάσεων. ούτω ώστε ε, στο μέλλον με τη συνεργασία να ε, μπορέσουν να κατασκευαστούν στο μέλλον ηλιακές ή αιωλικές εγκαταστάσεις θαλάσσιες Και στο πλαίσιο αυτή της συνεργασία, ε, ε, αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μας βοηθήσουν στην υλοποίηση του μηχανισμού συνδέοντα την Ευρώπη. Ε, άλλος τρόπος ε, συνεργασίας θα είναι ο μελλοντικό πληρωτικό μηχανισμός όπου μία χώρα υποδοχή θα μπορεί να παρέχει λειτουργία στατιστικής μεταφοράς για όσους ε, Υπηρεσίε ε, για όσου ε, δεν έχουν τόσο καλέ περιβαλλοντικέ συνθήκε. Αυτό ο μηχανισμό λειτουργεί ήδη πριν δύο χρόνια. Η Εστονία μαζί με τη Λουθανία ήταν μεταξύ των πρώτων που χρησιμοποίησαν αυτό το statistical transfer και μεταφέραμε και βοηθήσαμε το Λουξεμβούργο να εκπληρώσει του στόχου του. Ε, τώρα θεωρούμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε πιο προχωρημένο στάδιο. Επερώτηση, κύριε Πέτρεσαν. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την ε, άριστη απάντησή σας. Ε, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει χρηματοδότηση και ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το μηχανισμό που λέτε και να καταπολεμήσουμε ε, την κλιματική αλλαγή χρησιμοποιώντα περισσότερα θαλάσσια αιωλικά πάρκα. Πώς θα διασφαλίσετε εσεί ε, την απαραίτητη χρηματοδότηση. Αναφέρατε το μηχανισμό συνδέοντα στην Ευρώπη που αναφέραμε πριν από τις εκλογέ και είπαμε ότι το 50% θα αφιερωθεί στη διασυνορική συνεργασία και την ενέργεια. Τι θα κάνετε εσεί ε, σε θέματα περιφερειακή συνεργασία, όπω στη Βαλτική και στη Βορεια Θάλασσα. Πώς θα διασφαλίσετε ότι θα ληφθούν υπόψη για χρηματοδότηση. Επίσης θα ήθελα να ε, απαντήσετε και στην άλλη ερώτηση που έκανε ο κ. Βιούσεκ για το δάνειο. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να βοηθηθούμε έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και να προωθήσουμε την ανάπτυξη, την πράσινη ανάπτυξη. Ευχαριστώ κ. Σίμψον. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα μελλοντικά έργα τέτοιου τύπου χρειάζονται διαφορετική χρηματοδότηση, πιστεύω. Εν μέρη μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη, αλλά επειδή μπορεί να είναι μεγάλης κλίμακας, μπορεί να χρειαστεί και συγχρηματοδότηση είτε από ιδιωτικές τράπεζες, είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που εν μέρη θα μετατραπεί σε κλιματική τράπεζα. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, η τεχνολογία είναι φθηνότερη πλέον ε, σε σχέση με πριν από 10 χρόνια και μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστική ε, όσον αφορά τις τιμές της αγοράς. Οπότε υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην χρειαστούν επιπλέον μηχανισμούς υποστήριξης. Αυτό το παράθυρο για τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας έχει σχεδιαστεί και δημιουργηθεί ειδικά για την πρόθεση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των διαφορών κρατών μελών ούτως ώστε να μην επενδύει ο καθένας μας μόνος του στη δική του ε, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Είναι σοφότερο να το κάνουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι ο κ. Μενίστο που εκπροσωπεί τους Πρασίνους. Ε, ε Σίτρα. Κυρία Πρόεδρε, το κλίμα είναι η πιο σημαντική πρόκληση και η υπαρξιακή απειλή που έχουμε να χειριστούμε στη δική μας ε, διάρκεια ζωής. Και εσείς είπατε ότι θα επιτύχουμε τους στόχους ε, απαλλαγή από τον άνθρακα μέχρι το 2050 και θα είμαστε επίσης σε πάνω από τους στόχους για το 2030. Αυτό είναι πολύ καλά. Το κόμμα σας όμως ε, αρνήθηκε να βάλει στην πολιτική για την πάυση του άνθρακα το 2050 όταν εσείς υπηρετούσατε. Επίσης γνωρίζουμε ότι έχετε στηρίξει την ε, πετρελαιοβιομηχανία στη χώρα σας. Η αισθανική κυβέρνηση τώρα ε, θέλει να επενδύσει δε στη πετρέλαιο. Και επίση, ε, ε, κατά τη διάρκεια τη δική σα θητεία ε, συνεχίσατε τι επιδοτήσει στα παραδοσιακά, στους παραδοσιακούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Πώς λοιπόν δεσμεύεστε να πάψει η χρήση των ορυκτών καυσίμων και πώ θα δείξετε ότι εσεί προσωπικά είστε προσιλωμένοι στην επίτευξη αυτών των στόχων. Σα ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Κοιτάξτε, όπω ανέφερα στι ενορυκτήριές μου παρατηρήσει διατέλεσα υπουργό ε, Ενέργεια ε, στην Εστονική Κυβέρνηση και στη διάρκεια εκείνη τη περίοδου υιοθετήσαμε ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα για την ενέργεια ε, πρόγραμμα δράσης για την ενέργεια, σύμφωνα με το οποίο οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα μειωνόταν 70% μέχρι το 2030. Παράλληλα, είχαμε ένα μακροχρόνιο, μακροπρόθεσμο μάλλον πρόγραμμα για το κλίμα που θέσπιζε την μείωση των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050. 180%. Αυτά πριν δύο χρόνια και ήταν πολύ φιλόδοξα. Είναι αλήθεια ότι στις αρχές ε, της φετινής χρονιάς είχαμε λάβαμε αποφάσεις κοινοβουλευτικές, όμως μέχρι τώρα οι υπηρεσίες μας έχουν κάνει μια αξιολόγηση κινδύνου, γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει και πόσο θα κοστίσει ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στην κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Μάλιστα αυτή την εβδομάδα στην Εστονία αποφασίζεται και μάλλον συζητιέται το θέμα και στο επίπεδο το κυβερνητικό. Εγώ το, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαι προσιλωμένη 100% στην επίτευξη αυτού του στόχου. Πιστεύω πως η εστονική κυβέρνηση θα ανταποκριθεί και θα αποδώσει όπως ε, πέτυχε και τους στόχους του ε, τους ισχύοντες τους στόχους για το 2030, η Εστονία νίκη στην ομάδα πράσινης ανάπτυξης και ανέκαθεν ήταν φιλόδοξη με τους περιβαλλοντικούς στόχους. Επερώτηση. Σας ευχαριστώ για τη δέσμευσή σας γι' αυτό, αλλά δεν απαντήσατε στην ερώτηση για τις επιδοτήσει. Ε, ε, επίσης, όσον αφορά τους στόχους του 2030, η κυρία Βόντερ Λόιεν δεσμεύθηκε στην αύξηση των στόχων από 50% στο 55%, πράγμα το οποίο δεν είναι σύμμορφο προς τις φιλοδοξίες του Παρισιού. Πολλά πρέπει να γίνουν και όταν πρόκειται για τα ανανεώσι, τις ανανεώσιμες και την ε, ενεργειακή απόδοση, τα προγράμματα αυτά που ακολουθούνται δεν ανταποκρίνονται καν στους ισχύοντες στόχους. Πολλά πρέπει να γίνουν λοιπόν και για τις ανανεώσιμες. Ως κομμάτι του Green Deal θα πρέπει να είναι πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμα επενδύσεων στις ανανεώσιμες και στην ε, ενεργειακή απόδοση. Αυτό σημαίνει όμως αύξηση των στόχων για το 2030 και επίση και ότι η Κομισιόν θα αντιμετωπίσει το κενό ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς στόχους και τις φιλοδοξίες των κρατών μελών. Πώς ε, θα ανταποκριθείτε σε αυτά όλα με συγκεκριμένα μέτρα. Δεν δώσατε συγκεκριμένα μέτρα στις γραπτές σας απαντήσεις. Ναι, ευχαριστώ και θα επανέλθω στην πρώτη για το σχιστολιθικό πετρέλαιο. Ε, μάλιστα, για το, το, το ETS λειτουργεί η ανταλλαγή, το εμπόριο μάλλον εκπομπών. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς η παραγωγή ενέργειας από το σχιστολιθικό πετρελαίο μειώνεται. Ε, εισάγουμε αντί αυτού ε, σκανδιναβική ενέργεια από τη Φιλανδία, πυρηνική παραγωγής και αντικαθιστούμε και με ανανεώσιμες για την επίτευξη των στόχων εάν εφαρμοστεί πλήρως το δίκτυο και λειτουργήσει, τότε ο τομέας ενεργειακός θα αποδώσει και θα καταφέρει τους στόχους που έχουμε ήδη υποσχεθεί και μετά θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τους στόχους. Αυτό που υποσχέθηκε δηλαδή η υποψήφια πρόεδρος 50% και προς 55%. Εγώ δεσμεύομαι για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ε, ο κ. Μπουχάιτ. Καλημέρα σας κύριε Σίμψον. Εδώ είμαι. Στη μέση. Κύριε Σίμψον, με ένα πρόγραμμα δράσης για τη χρηματοδότηση ε, της αηφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης. Εξήγηλε ε, νέα χρηματοδότηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, το Μάρτιο του 2018. και η πρωτοβουλία ήρθε το Μάρτιο του 2019 εδώ σε πρώτη ανάγνωση. Αυτό θα οδηγήσει σε σχεδιαζόμενη οικονομία και στρεβλώσεις στην αγορά. Ιδιαίτερα ο ιδιωτικός τομέας θα πάρει τη μερίδα του Λέοντος 180 ε, δισεκατομμύρια ε, για να εφαρμοστεί αυτή η ε, πολιτική ετησίως. Αυτό πώς το αξιολογείτε. Καλείται η ευρωπαϊκή ιδιωτική οικονομία να χρηματοδοτήσει μια ιδεολογική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πατάει κατάφορα την ελεύθερη οικονομία της αγοράς και ε, τον απρόσκοπτο ανταγωνισμό. Ε, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Για τους κλιματικούς μας στόχους πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει πώς να το πω να συνεισφέρουν και ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να εποφεληθεί από τη σταδιακή εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων. Και θα εποφεληθεί από την έρευνα και την καινοτομία στο μέλλον. Αν θέλει η Ευρώπη να είναι ηγέτης σε αυτή την προσπάθεια, χρειάζεται μεγαλύτερη καινοτομία Έτσι θα έχουμε περισσότερες εργασίες, περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερη ανταγωνιστικότητα. Ταυτόχρονα έχουμε δεσμευτεί για κάποιους στόχους σε σχέση με το κλίμα και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι αυτό θα γίνει με τρόπο ε, που να συμφέρει. Να είναι ασφαλείς οι ενεργειακές πηγές μας, να μην απειλείται δηλαδή η ενεργειακή ασφάλεια αλλά και ταυτόχρονα οι τιμές να παραμένουν προσιτές. Δεν είναι δυνατό να αυξηθούν τα τιμολόγια δραματικά. Και αν εξασφαλίσουμε αυτές τις βασικές λοιπόν υποθέσεις που κάνουμε και παραδοχές, τότε μπορώ να πω ότι ε, είναι εφικτό να φτάσουμε να πιάσουμε τους στόχους που έχουμε για το κλίμα. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση. Ο κύριος Μποχάιτ. Δεν απαντήσατε ακριβώς αυτό που σας ρώτησα, να το πω πιο συγκεκριμένα. Το θέμα είναι εξής. Δεν είναι ότι δεν θα επωφεληθεί η ιδιωτική οικονομία δεν είναι δεδομένο κάθε στιγμή. Αλλά στο πακέτο αυτό ή σε άλλα έχετε προβλέψει μέτρα για την υποστήριξη της βιομηχανίας μας, ε, ε, η οποία βρίσκεται μπροστά σε ένα κατακλυσμό. Γίνονται βαθιές αλλαγές και αυξάνεται ε, αυτή η πρόκληση όλο και περισσότερο. Απάντησε. Αυτό είναι ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Uh, Θα πρέπει οι ενεργειακές τιμές ε, να είναι ε, ανταγωνιστικές. Η τιμολόγηση της ενέργειας δηλαδή. Και να μπορούμε να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις στα δίκτυα. μην είναι όλες οι επενδύσεις για τους καταναλωτές, ας πούμε. Να ανοίξει η αγορά, να είναι ανταγωνιστική με πολλούς παρόχους. Και έτσι οι τιμές θα είναι φθηνότερες. Οι τελικές τιμές του καταναλωτή. Και αν οι αγορές μας είναι διασυνδεδεμένες, που δεν είναι ακόμα, γιατί υπάρχουν ακόμα προβλήματα και ε, λείπουν και οι κρίκοι για να συνδεθούν όλα τα δίκτυα, τότε θα δίνουμε ε, σε μεγαλύτερες αγορές ανανεώσιμες. Αυτός ήταν και ο βασικός στόχος του ενεργειακού πακέτου, του πράσινου ενεργειακού πακέτου. Ότι στο κέντρο της αγοράς θα είναι οι καταναλωτές και η τιμή θα μείνει προσιτή. Ευχαριστώ. Thank you very much. Um, now, the next is... Ευχαριστούμε. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κρασνατέψκι από το ECR. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, στο πρόσφατο ψηφισμά του για την ε, αγωγό φυσικό αέριο ΟΠΑΛΑ το δικαστήριο αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην απόφασή του στην αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης. Αυτή η ενεργειακή αλληλεγγύη και η ενεργειακή ασφάλεια θεσπίζεται όπως ξέρουμε στο άρθρο 194 της συνθήκης ε, της, Ευρωπαϊκής, της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά την περαιτέρω εφαρμογή αυτής της αρχής. Ως μελλοντική επίτροπος θα υποστηρίξετε την ιδέα των υποχρεωτικών stress test για να ελέγχεται η ενεργειακή ασφάλεια και αυτό να εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε εγκατάσταση ε, ενεργειακής υποδομής. Ε, θα ε, χρησιμοποιήσετε νέα κριτήρια και δείκτες που θα μας βοηθούν να αξιολογούμε κατά πόσο τηρείται πραγματικά η αρχή της ενεργειακής αλληλεγγύης και ασφάλειας. Η Επιτροπή θα προτείνει σαφή κριτήρια αξιολόγησης του πότε υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις για την ασφάλεια, για την ενεργειακή ασφάλεια και την ασφάλεια ευωδιασμού, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της οδηγίας για το φυσικό αέριο. ευχαριστώ κύριε Κρασνοδεύσκη, για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο του φυσικού αερίου. Βλέπουμε με ύψιστη σοβαρότητα την πτύχη της αλληλεγγύης. Όπως υπόθηκε πολύ σωστά σε αυτή την υπόθεση, έχουμε αυτή την απόφαση του δικαστηρίου που ε, βάσει της οποίας πρέπει να έχουμε στο νου μας και την πτυχή της αλληλεγγύης. Πιστεύω ότι όταν αναφερόμαστε στην σύνθεση που θα έχει η μελλοντική αγορά φυσικού αερίου, αυτός θα είναι ο βασικός πυλώνας. Όσαν, όταν μιλάμε για το φυσικό αέριο δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο σημαντική είναι η διαφυροποίηση των ε, πηγών. Από αυτή την άποψη η Πολωνία, η χώρα από την οποία εσείς προέρχεστε, έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Έχετε ένα τερματικό LNG, έχετε σύνδεση με τη Λιθουανία, θα έχετε έναν αγωγό φυσικού αερίου προς την Νορβηγία, τρεις διαφορετικές πηγές. Κατάσταση αξιοζήλευτη για πολλές άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ. Still have time if you wish. You still have time if you wish. Uh, uh, Mr. Krasnodebski, you want to put a follow-up question? Okay, follow-up question. Κύριε Κρασνοδεύσκη, έχετε επερώτηση λίγο πιο γενικά. Αφού μιλάμε για αυτή την πολύ σημαντική μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την συνοχή, τη συνέπεια της μετάβασης σε τέτοιου είδους οικονομία βάσει της αρχής της ε, τεχνολογικής ουδετερότητας που ε, θεσπίζεται από τις συνθήκες ε, και που αποδίδει σε κάθε κράτος μέλος την ευθύνη του να καθορίσει μόνο του το ενεργειακό του μείγμα. Ευχαριστούμε κυρία Σίμψον. Αν κατάλαβα καλά την επερώτηση, Ρωτήσατε για τις μελλοντικέ προοπτικές ε, των επενδύσεων σε φυσικό αέριο. Ναι, σωστά. Πράγματι, το ενεργειακό μείγμα αποφασίζεται καθαρά από κάθε κράτος μέλος για το ίδιο το κράτος μέλος. Και ξέρετε, σε αυτή τη μεταβατική περίοδο το ποσοστό του φυσικού αερίου ως ε, πηγής ενέργειας ε, δεν θα μειωθεί σημαντικά. Ε, μάλλον θα αυξηθεί σημαντικά γιατί πολλές χώρες θα αντικαταστήσουν τον άνθρακα με φυσικό αέριο. Αλλά ταυτόχρονα όταν μιλάμε για μελλοντικές επενδύσεις δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι επενδύσεις αυτές στα δίκτυα φυσικού αερίου θα πρέπει να αποδώσουν και στο μέλλον. Και λέγοντας κάτι τέτοιο εννοώ ότι Υπάρχουν και άλλα αέρια πέραν του φυσικού αερίου που έχουν μικρότερο ε, περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στο ε, υδρογόνο, στα βιοαέρια. Τα δίκτυα αυτά θα πρέπει να έχουν αποδοτικότητα και στο μέλλον, δηλαδή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μετά το 2030. αλλά κατά τη μεταβατική περίοδο, μάλλον μέχρι τη μεταβατική περίοδο, τα, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν τα δίκτυα φυσικού αερίου και οι διασυνδέσει. Ευχαριστούμε. Ο επόμενο μιλητής είναι ο κύριος Μποτέγκα από την ΚΟΕ. Oui, Μάλιστα, καλημέρα σας, ευχαριστώ. Εγώ πρέπει να μπω κάπως σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ, εδώ πίσω είμαι. Στην επιστολή περί της εντολής σας, η κυρία Βαντελαΐεν σας ε, λέει να αποκομίσετε όλο το δυναμικό του υγροποιημένου ε, φυσικού αερίου. Το είπατε και εσείς πριν από λίγο. Θα είμαι λοιπόν πολύ συγκεκριμένος. Ποια μέτρα προβλέπετε. Ε, αυτό σημαίνει πως θα επενδύσετε στις υποδομές φυσικού αερίου. θα τοποθείτε στηθείτε οικονομικά πολύ ξεκάθαρα σε αυτήν την ε, ε, γραμμή και σε σχέση με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας ε, στην οποία θα συμβάλλετε. Είναι η οδηγία που ορίζει το μίνιμουμ φορολόγησης για τα καύσιμα και για τον ηλεκτρισμό. Τι θα κάνετε για να μειώσετε τις, εκπομπές, σε ποιο καύσιμο θα στοχεύσετε. Σα ευχαριστώ η κυρία Σίμψον. Μάλιστα, όντω. Υπάρχει μια παράγραφος στην επιστολή της εντολής μου για την πρόθεση του υγροποιημένου ε, φυσικού αερίου και εγώ το θεωρώ ότι θα συμβάλλει αυτό στην ασφάλεια γιατί η ασφάλεια ε, ανεφοδιασμού θα προκύψει από τη διαφοροποίηση των πηγών και αυτό σημαίνει πως θα υπάρξουν επενδύσεις ε, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Γίνονται επενδύσεις αυτή τη στιγμή, είναι υπό εξέλιξη στην Κροατία και επίσης στην Βαλτική θάλασσα και στην Πολωνία. Όσον αφορά τη φορολογία των, α, ε, της ενέργειας, αναφέρεται αυτό και στη δική μου εντολή. Θα συνεργαστώ στενά με τον Επίτροπο Τζεντιλόνη. Ε, γι' αυτό είναι αλήθεια ότι αυτή η οδηγία είναι ήδη χρονολογείται εδώ και 15 χρόνια. Οπότε δεν μας βοηθά όσο θα μπορούσε στο να επιτύχουμε τους στόχους, τους ενεργειακούς και τους κλιματικούς και δεν πιστεύω πως... Ε, πιστεύω μάλλον ότι η δυσκολία είναι ότι επιτρέπει εξαιρέσεις για τα ορυκτά καύσιμα. Πράγμα που καθιστά δύσκολη τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα ορυκτά καύσιμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα, αν με ρωτάτε τι είδους φορολογία θα προτείνω, βεβαίως αυτό θα είναι σύμφωνα με τους ενεργειακούς και κλιματικούς μας στόχους. και θα είναι προς την ε, προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ανανεώσιμων. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Επερώτηση. Κύριε Ποτέγκα. Μάλιστα. Ακούγοντάς σας φοβούμε πως το μήνυμα το οποίο στηρίζουν οι νέοι για το κλίμα και τα κίτρινα γυλαίκα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχει ακουστεί ακριβώς. Είναι σαφές ότι αν έχουμε ένα Έχουμε τους νέους που ζητούν ε, επενδύσεις στην ανανεώσιμη ενέργεια, ένα ευρώ που έχουμε δεν μπορούμε να το επενδύσουμε και για τα καύσιμα που συνεχίζουν να ρηπαίνουν και για τις ανανεώσιμες. Εγώ θέλω να ακούσω μια σαφή δέσμευση υπέρ των ανανεώσιμων και εις βάρος των ε, ε, ρηπογόνων ενεργειών. Και ποιος θα τα πληρώσει αυτά, γιατί εγώ φοβούμαι πως οι εργαζόμενοι θα χρειαστεί να πληρώσουν την ύφη και όχι μεγάλες πολυεθνικές θα μας εγγυηθείτε ότι δεν θα βαρύνουν όλα αυτά τον κόσμο. Ευχαριστώ κύριε Ποτέγκα. Μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι το μήνυμα των νέων έχει πολύ εισακουστεί και το πρόγραμμα δράσης ε, που θα ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες ε, θα το δείτε. Χρειάζεται όντω επενδύσει στι ανανεώσιμε. Υπάρχουν διάφορες βάσει ε, βάσεις επί των οποίων θα στηριχθούμε. Ε, μία από αυτές είναι τα κονδύλια ε, τα ευρωπαϊκά, το Horizon Europe, το LIFE και άλλα. Άλλη επιλογή είναι ο δανεισμός με ιδιωτικό χρήμα Θα έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο, πράγμα που είναι αρμοδιότητα του Αντιπροέδρου Ντομπρόφσκης και για τις μελλοντικέ επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Πάντως, εν γέννη, και μέσα στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα δοθούν περισσότερα χρήματα στην έρευνα και στην ανάπτυξη από ό,τι στο προηγούμενο για την ενέργεια. Η Πρόεδρος, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Ας προσπαθήσουμε να τηρούμε το χρόνο μας όπως συμφωνήσαμε αρχικά. Αρχίζει τώρα ο δεύτερος γύρος των ομιλιών. Ο κύριος Γκιούρκ πρώτος ε, από την Επιτροπή Ήτρα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Thank you, Commissioner Ευχαριστώ, κυρία Υποψήφια Επίτροπη. Ε, συμμεριζόμαστε όλοι τις φιλοδοξίες σας για την κλιματική ουδετερότητα, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εξαρτάται από την υποστήριξη του κόσμου, των πολιτών για να πετύχουμε θα πρέπει να τους εξασφαλίσουμε, να τους καθησυχάσουμε και θα πρέπει να έχουν καλή ενημέρωση ότι δεν θα κινδυνεύσουν να μείνουν πίσω. Ε, θέλω να σας ρωτήσω συγκεκριμένα. Έχετε ποσοτικοποιημένες αναλύσεις και πότε θα τις φέρετε για το εφικτό του στόχου 2050. Πόσο χρόνο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τα μελετήσει όλα αυτά για να μην μείνει κανένας πίσω και καμία ε, περιφέρεια. Και πώς ε, θα εγγυηθείτε ότι δεν θα εκραγούν οι τιμές και δεν θα δικημευτεί ο εφοδιασμός της ασφάλειας της ενέργειας στα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Kirk, for your question. And, uh, indeed... Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πραγματικά αυτό είναι μεγάλη ανησυχία πολλών ευρωβουλευτών και φυσικά και κρατών μελών το κόστος της μετάφασης δηλαδή και ποιος θα το πληρώσει. Θα πρέπει να είναι δίκαιο, ιδιαίτερα όταν έχουμε υπόψη ότι τα κράτη-μέλη δεν ξεκινούν όλα από την ίδια φετηρία. Υπάρχουν κάποια κράτη που ακόμα εξαρτώνται από τα ορυκτά καύσιμα και κάποια άλλα τα οποία βρίσκονται σε πιο προηγμένο στάδιο. Με ρωτήσατε το συγκεκριμένο σχέδιο για τους στόχους του 2050. Μπορώ να σας πω το εξής. Θα συνεργαστώ στενά με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Φρανς Τίμερμανς, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος επίτροπος για την κλιματική νομοθεσία. Πριν γίνουν όλα αυτά, πρέπει να μελετηθεί σε βάθος ο αντίκτυπος και να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς θα φτάσουμε στους στόχους του 2050. Μέχρι το 2021 να έχει καταρτιστεί αυτό το σχέδιο. Εγώ ως αρμόδια για την ενέργεια ε, θα πρέπει να εξασφαλίσω ότι παράλληλα με αυτή την ε, φιλόδοξη ε, νομοθεσία για το κλίμα ε, θα πρέπει να φροντίσω να εξασφαλίσω ε, τους καταναλωτές και τις εταιρείες μας. Να είναι η ενέργεια προσιτή και ανταγωνιστική. Για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει να επενδύσουμε στα ενεργειακά μας δίκτυα, αλλά και ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε το υπάρχον πλαίσιο. Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω για την εσωτερική αγορά και τα ωφέλη της. Ελπίζω στη συνέχεια να μου δοθεί ευκαιρία. Ε, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ. Αναφέρατε την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας στις απαντήσεις σας και εδώ και στις γραπτές σας στο ερωτηματολόγιο και συμφωνώ. Και ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι στην κεντρική Ευρώπη Χρειάζεται οπωσδήποτε πυρηνική ενέργεια για να ξεφύγουμε από τον άνθρακα και να είναι προστατευμένοι και οι πολίτες από τους κινδύνους και των τιμολογίων και του ενεφοδιασμού. Χωρίς αυτά θα είναι πιο ακριβή η ενεργειακή μετάβαση στο νέο σχέδιό σας για τις βιώσιμες επενδύσεις, τι χώρο σκοπεύετε να δώσετε και τι θέση στην πυρηνική ενέργεια. Ευχαριστώ. Η πυρηνική ενέργεια θα είναι τμήμα ε, του ε, ενεργειακού μείγματος. Αυτό το αποφασίζει κάθε κράτος μέλος. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε χώρες οι οποίες κλείνουν τα πυρηνικά τους εργοστάσια σιγά σιγά και κάποια άλλα κράτη-μέλη σχεδιάζουν να χτίσουν καινούργια για να κλείσουν τα ε, θερμοηλεκτρικά εργοστάσια ε, από άνθρακα δηλαδή. Η Φιλανδία μόλις εγκαινίασε ένα νέο πυρηνικό εργοστάσιο. Αυτό είναι απόφαση του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά πώς διαμορφώνει το ενεργειακό μείγμα και από ποιες πηγές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμείς ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι είναι ακριβώ ασφαλή τα πυρηνικά εργοστάσια και η διαχείριση των αποβλήτων είναι ασφαλής για το περιβάλλον. Όχι μόνο εντός Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην άμεση γειτονία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Φούγκλσανκ, Σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Εδώ είμαι, στην πρώτη σειρά. Κυρία Υποψήφια Επίτροπη, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θέλω να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο αυτό που θα ρωτήσω. Γιατί τους στόχους ανανεώσιμων, σύμφωνα με τις γραπτές σας απαντήσεις, θα εκτιμήσετε αν χρειάζεται αναθεώρηση η κείμενη νομοθεσία για τα ενεργειακά για να φτάσουμε στο στόχο ε, της μείωσης κατά 55% των ρήπων μέχρι το 2030. Συμφωνεί η υποψήφια επίτροπος με τους διάφορους εμπειρογνώμονες και ΜΚΟ που λέγουν ότι χρειαζόμαστε πολύ υψηλότερους στόχους, πολύ υψηλότερους στόχους από ότι το 32% ανανεώσιμων μέχρι το 2030. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες ανανεώσιμες ε, που να φτάνουν μέχρι το 45% του ενεργειακού μείγματος. Συμφωνεί η υποψήφια επίτροπος με αυτή την παραδοχή. Ευχαριστώ κύριε Φόγγελσανγκ για τις ανανεώσιμες. Υπάρχουν κάποιοι στόχοι για το 2030, τους οποίους διαπραγματευτήκαμε. Και τώρα βρισκόμαστε στην κατάσταση μετά από ένα τρίμηνο, μέχρι το τέλος του έτους, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δώσουν ε, τα πρώτα σχέδια, τα εθνικά του σχέδια για την εφαρμογή όλων αυτών. Για να μας δώσουν όμως συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς σκοπεύουν να φτάσουν στους στόχους τους. παρά το γεγονός ότι πολλά κράτη-μέλη ακόμα καταρτίζουν αυτά τα σχέδια για να φτάσουν σε αυτούς τους υποστόχους. Πολλά έχουν υποσχεθεί ότι θα αυξήσουν το ποσοστό. Την περασμένη Τρίτη συνεδρίασε το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας και διάφορες χώρες ανακοίνωσαν ότι σε κρατικό επίπεδο ήδη είχαν λάβει αποφάσεις να στοχεύσουν υψηλότερα ποσοστά από τα συμπεφωνημένα στο πακέτο για την καθαρή ενέργεια. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και εκείνα τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ευνοϊκές περιβαλλοντικές ε, συνθήκες να συνεργαστούν με άλλους για να φτάσουν στους στόχους. Και αυτός ο μηχανισμός συνεργασίας θα δημιουργηθεί. Ευχαριστώ. Επερώτηση κύριε Φούγκλτζανγκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που τα κράτη-μέλη αναθεωρούν τους στόχους και μάλιστα προς τα πάνω. Δεν είμαι βέβαιος ότι μου απαντήσατε αν συμφωνείτε εσείς ότι πρέπει να αυξηθούν οι στόχοι από το 32% στο 45% ή μέχρι και 45% μέχρι το 2030. Και αν ναι, θα την οδηγία για τις ανανεώσιμες με υψηλότερο αριθμητικό στόχο. Ναι ή όχι, αυτή είναι η απάντηση που περίμενα. Εγώ είμαι από την Εστονία. Δικός μας στόχος ε, είναι να έχουμε το 32% μέχρι το 2020 και μέχρι το 30 θα είμαστε στο 42-43%. Νομίζω ότι είναι εφικτό να στοχεύει κανείς σε ψηλότερα ποσοστά. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για τις ανανεώσιμες, για να εδρεωθούν. Ε, ας πούμε, να ερευνήσουμε, να δώσουμε κονδύλια στην έρευνα και την καινοτομία για την αποθήκευση. Ε, ανανεώσιμων. Και σε τοπικό επίπεδο πρώτα να δημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά τοπική για να μπορούν να φτάνουν σε ευρύτερες αγορές οι ανανεώσιμες και αυτές οι δράσεις είναι πολύ σημαντικές. Επίσης, θα επανέλθω σε αυτό το μηχανισμό συνεργασίας. Θα πρέπει να βοηθήσουμε έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να επενδύουν σε πάρκα, είτε είναι θαλάσσια αιωλικά πάρκα, ε, είτε είναι ηλιακά πάρκα κτλ. Ευχαριστώ. Φωτοβολταϊκά δηλαδή. Η κυρία Γκαμόν από την ομάδα Renew Europe. Thank you very much uh, for the strong commitment that um, σας ευχαριστώ πολύ για τις δεσμεύσεις που μας ε, έχετε κάνει στις γραπτές σας απαντήσεις αλλά και σήμερα για την επίτευξη των κλιματικών στόχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς στο Renew Europe πιστεύουμε πως πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς αλλά πρέπει αυτό να γίνει και εγκαίρως διότι ο χρόνος ε, τελειώνει. Εσείς θα είστε επικεφαλής αυτών των προσπαθειών ιδιαίτερα όσον αφορά τη διευκόλυνση των project ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η Ενέργειες είναι ας πούμε η υδροελεκτρική ενέργεια ή η αιωλική ενέργεια, οι οποίε υπόκειται σε διάφορα άλλα ρυθμιστικά πλαίσια όπου και άλλοι επίτροποι είναι συνυπεύθυνοι. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε να αποδεσμεύσετε το πλήρες ε, δυναμικό που έχουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την υδροελεκτρική ενέργεια και την ε, αιωλική ενέργεια, ώστε να λειτουργήσουν δηλαδή όλα αυτά τα προγράμματα ε, να είναι ευφυή, ε, ε, συνδυασμένα και αποδοτικά. Πώς μπορούμε αυτά περαιτέρω να τους δώσουμε και άλλη έμφαση. Κυρία Σίμψον, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Μάλιστα, χρειαζόμαστε περισσότερες ε, ε, εγκαταστάσεις για τις ανανεώσιμες για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και αυτό το χρειαζόμαστε, ε, χρειαζόμαστε και περισσότερες επενδύσεις εφόσον θέλουμε να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ε, υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχουν... Ε, προγράμματα με δημόσια αποδοχή αποδοχή μάλλον από τον ε, κόσμο, αλλά υπάρχουν και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και που πρέπει να κάνουμε ας πούμε, για τον προγραμματισμό, για τον σχεδιασμό, ζητάμε από τα κρατη ε, με βάση την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές, να ε, μπορέσουν να απλοποιήσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης ώστε να μην χρειάζεται, να μην είναι τόσο χρονοβόρες οι διαδικασίες πριν από, τα, από τις, ε, την υλοποίηση των επενδύσεων. Βεβαίως υπάρχουν και όρια, περιορισμοί. Πρέπει δηλαδή να δουλέψουμε στενά σε συνεργασία με τους επιτρόπους που είναι υπεύθυνοι ας πούμε για τη χρήση των γεών ή μιλάμε για ανανεώσιμες που προέρχονται από υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Εκεί θα πρέπει να συνεργαστώ με τον αρμόδιο επίτροπο ε, της ε, αλληλείας, αλλά Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, υπάρχουν ε, συγκεκριμένα προγράμματα. προσαρμοσμένα ε, και τα οποία θα προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Ε, βέβαια φαντάζομαι συναισθάνεστε την ευθύνη του συντονισμού όλων αυτών των προσπαθειών. Τι θα κάνετε για να βοηθήσετε τα κράτη-μέλη να ε, επιτύχουν και να ε, οικοδομήσουν αυτά τους τα προγράμματα εγκαίρως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να επιτύχουμε τους κλιματικούς στόχους. Όπως αναφέρατε, κάποια από αυτά τα προγράμματα αντιμετωπίζουν ε, ε, ε, καθυστερήσεις, πράγμα που κάνει δύσκολη την εφαρμογή των προγραμμάτων. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάθε κράτος μέλος να πετύχει τους στόχους. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι πολλοί από τους στόχους δεν έχουν επιτευχθεί ή έχουν καθυστερήσει. Για το 2020 υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους μπορεί να μην επιτευχθούν οι στόχοι των ανανεώσιμων. Ένας λόγος είναι ότι έχουν καθυστερήσει στην εφαρμογή τους κάποιες πρωτοβουλίες και ο άλλος είναι ότι τα μέτρα έχουν υπολογιστεί με εξαιρετικά θετικό τρόπο. Τώρα, λόγω της ε, συνεργασίας με τα κράτη-μέλη θα έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία για κάθε κράτος. Θα πάρουμε λοιπόν τις εκθέσεις για το τι έχει υλοποιηθεί και θα δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε ώστε να τους βοηθήσουμε όλους να τηρήσουν τις προθεσμίες. Οι εκθέσεις αυτές θα είναι διαθέσιμες και θα δοθούν και στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε την έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης και εκεί θα έχουμε και τις πληροφορίες και θα μεριμνούμε ώστε να μην καθυστερούν πρωτοβουλίες αυτές. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ε, μόνη ε, ε, μάλλον μόνος ε, έμβη, ε, από την ΕΜΔΙ, ο κύριος Πέτερ Λίζε. Θα ήθελα να επανέλθουμε στο ζήτημα της κλιματικής ουδετερότητας. Στη Σύνοδο Κορυφής η Εστονία ήταν κατά και αυτό είχε συνέπειες στην Νέα Υόρκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε να δεσμευτεί στην κλιματική ουδετερότητα και θέλω να καταλάβω τι ρόλο διαδραματίσατε εσείς προσωπικά. Εξηγήσατε δηλαδή τη θέση της κυβέρνησης, αλλά ποια ήταν η προσωπική σας θέση πριν από τη Σύνοδο του Ιουνίου. Αναφερθήκατε σε κάποια ανάλυση που χρειάστηκε να κάνει η κυβέρνησή σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεστε την ανάλυση του σημερινού Επιτρόπου Ενέργειας του κ. Κανιέτε. Διότι ήδη από τον Νοέμβριο η Κομισιόν έκανε ανάλυση και το ερώτημά μου είναι εσείς ως υπουργό δεν εμπιστευτήκατε την ανάλυση της Κομισιόν και να σας υπενθυμίσω ότι δεν απαντήσατε την απάντηση ε, του κυρίου Μπούζε και τη ρωσική ε, παρέμβαση για την υπόθεση του φυσικού αερίου. Ευχαριστούμε κυρία Σίμψον. Ευχαριστώ κύριε Λίζε. μετά από τις ε, κοινοβουλευτικές εκλογές ε, στην Ιστονία το Μάρτιο είμαι μέλος του Κοινοβουλίου. Δεν ήμουν τον αιώνιο πια υπουργό Ενέργειας, ήμουν μέλος του Ιστονικού Κοινοβουλίου. Όπως εξήγησα όμως νωρίτερα, η Εστονία ε, έχει υπάρξει ιδιαίτερα φιλόδοξη και αφοσιωμένη στα κλιματικά σχέδια. Πριν δύο χρόνια, προσαρμόζοντας ε, το μακροχρόνιο σχέδιο δράσης μας για το κλίμα, αξιολογήσαμε όλες τις δυνατότητες, τι μπορούμε να κάνουμε, πόσο θα κοστίσει και υιοθετήσαμε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο για το κλίμα. Για εκείνη την εποχή, για το 2017 πέρασε από το Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με την νομοθεσία μας, χρειαζόμαστε και απόφαση του Κοινοβουλίου για να αλλάξει. Διακρίσαμε ότι θα μειώναμε τα αερία θερμοκηπίου κατά 80%. Τώρα έχουν γίνει, έχει γίνει η εκτίμηση αντικτύπου και η σημερινή μας κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα κλιματικό συμβούλιο με 7 ε, υπουργούς κλειδί που είναι μέλη αυτού του Κλιματικού Συμβουλίου όπου συζητείται αυτό το ενδεχόμενο ε, της κλιματικής ουδετερότητας ε, αυτή την εβδομάδα. Από όσο γνωρίζω υπάρχει ένα σχέδιο δράσης για την επίδευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Μέχρι το Δεκέμβριο, όταν θα αποφασίσει σχετικά το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω ότι θα υπάρξει ομοφωνία Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να υποφεληθούν όλα τα κράτη-μέλη. Αν η Ευρώπη ηγηθεί στο μέτωπο αυτό. Ε, επερώτηση. Ευχαριστούμε για την απάντησή σας, αλλά δεν απαντήσατε την ερώτηση ποια ήταν η προσωπική σας θέση. Δεν ήσασταν υπουργό, αλλά ήσασταν ε, βουλευτής έγινε η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το παρόν κοινοβούλιο είπε ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να δεσμευτεί ε, για την κλιματική ουδετερότητα ήδη από τον Μάιο και τον Ιούνιο η Εστονία εξακολουθούσε να είναι κατά. Εσείς υποστηρίζετε δηλαδή την ιδέα, υποστηρίξετε την ιδέα της κλιματικής ουδετερότητας εσείς ως βουλευτής ή ήσασταν μέλος μιας πλειοψηφίας που είπε η Εστονία δεν μπορεί να δεσμευτεί. Κυρία Σίμψον. Από όσο γνωρίζω, η ερώτηση αυτή δεν εμφανίστηκε στην Ολομέλεια του Ιστονικού Κοινοβουλίου. Με αυτήν ασχολήθηκε μια ειδική επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων. Η θέση της Εστονίας δεν ήταν κατά. Απλά η Εστονία χρειαζόταν λίγο περισσότερο χρόνο για διαδικαστικούς λόγους Θέλαμε να κάνουμε μια αξιολόγηση του τι θα κάνουμε για να είμαστε έτοιμοι, για να είμαστε κλιματικά ουδέτεροι μέχρι το 2050. Και τώρα, αν μα συγκρίνετε με άλλε χώρε, πιστεύω ότι ήδη βρισκόμαστε μπροστά. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε και ένα από αυτά τα πράγματα είναι ότι η παραγωγή μας χιστολιθικού πετρελαίου ε, σε μια ιδιαίτερη περιοχή στην Εστονία, γίνεται αυτό σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ε, υφίσταται τεράστιες αλλαγές. Αν θέλετε να σας αναφέρω τη δική μου προσωπική δέσμευση, εγώ ναι υποστηρίζω την κλιματική ουδετερότητα. Είναι αναγκαία για να επιτύχουμε αυτή τη μείωση του 1,5 βαθμού Κελσίου. Και για να καταλήξω κατά τη δική μου θητεία στο Ιστονικό Κοινοβούλιο, δεν έγινε τέτοια ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Next speaker is... Uh, Ευχαριστώ. Η κυρία Κουταχάρ, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Η κυρία Σίμψον. Οι πρόσφατες επιθέσεις στα δηληστήρια στη Σαουδική Αραβία έδειξαν πόσο ευαίσθητη ε, είναι η ισορροπία και πόσο εύθραυστη ε, ε, είναι αυτή η ισορροπία του εφοδιασμού. Έγιναν πολλά για να διαφοροποιηθεί ο εφοδιασμός από τρίτες χώρες με υγροποιημένο φυσικό αέριο. Παρ' όλα αυτά ε, παραμένουμε εξαρτημένοι από μεγάλους παραγωγούς φυσικού αερίου όπως είναι η Ρωσία. Και όσο αυξάνονται οι κρίσεις στη Μέση Ανατολή μπορεί να αυξηθεί η δική μας εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Θα πρέπει λοιπόν να μειωθεί η ε, ε, εξάρτηση και να διαφοροποιήσουμε τις πηγές μας. Αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για άλλα στοιχεία της Ενεργειακής Ένωσης, ιδιαίτερα για τον γενικό μας στόχο να έχουμε μια οικονομία ουδέτερη ως προς τον άνθρακα. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που θα προτείνετε κατά τη διάρκεια της θητείας σας, έτσι ώστε η ασφάλεια του εφοδιασμού να είναι συμβατή με άλλα ζητήματα, όπως η απαγκίστρωση και επεξάρτηση από το διοξίδιο του άνθρακα. Ευχαριστώ. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Είναι γεγονός ότι η Ευρώπη ε, ήταν πάρα πολύ εξαρτημένη από εισαγωγές ενέργειας. and Έχουμε, ε, ε, εισάγουμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο Και αυτό θα παραμείνει και κατά τη μεταβατική περίοδο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής. Είναι βασική αρχή μας η ενέργεια να προέρχεται από ασφαλείς πηγές και να προστατεύουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια. Για το λόγο αυτό πρέπει να διαφοροποιήσουμε και τις πηγές μας, ε, προμήθευτές δηλαδή, αλλά και τις οδούς τις ενεργειακές. Ρωτήσατε για τις επενδύσεις στις ε, υποδομές φυσικού αερίου και χρειαζόμαστε επενδύσεις ε, και στις ανανεώσιμες. Κάποιες από τις επενδύσεις για τους αγωγούς φυσικού ανεργείου και τους θερματικούς σταθμούς ε, είναι βασικό στοιχείο της ενεργειακής μας ασφάλειας. Υπάρχουν και κάποιες διαδρομές ε, κάποια αγωγή που συγκεντρώνονται στη Βαλτική θάλασσα. Και οι βασικοί προμηθευτές έχουν μεγαλύτερο μερίδιο. Αλλά αυτό δεν συνάδει με την ενεργειακή μας πολιτική. Ε, συμπληρωματική ερώτηση. εκτός από την εξασφάλιση ότι δεν θα εξαρτώμαστε από κάποιες πηγές, σας ρώτησα και συγκεκριμένα τι μέτρα θα φέρετε για τις άλλες διαστάσεις όπως είναι η ε, απεξάρτηση από το διοξίδιο του άνθρακα των ενεργειακών μας συστημάτων. Και θέλω να σας ξαναρωτήσω γιατί υπάρχουν και νέες ε, απειλές, σύγχρονες, πέρα από την κλασική εξάρτηση, όπως είναι η κυβερνοασφάλεια και άλλες υποδομές που μπορεί να είναι ευάλωτες. Πώς θα τα αντιμετωπίσετε αυτά, είναι προτεραιότητά σας. Και σε 20 χρόνια ή μετά από 20 χρόνια όταν έρθουν οι Ευρωπαίοι να δουν τον απολογισμό σας, ποια θα είναι η κληρονομιά που θα έχετε αφήσει μετά από 5 χρόνια στην ενεργειακή ασφάλεια. Um, we have to, um, Um, Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας um, ότι υπάρχουν ε, διάφορες πηγές ενέργειας. Ε, αυτά όμως δεν είναι δωρεάν όλα. Έχουν κάποιο κόστος. Πρέπει να γίνουν κάποιες επενδύσεις. Ιδιαίτερα στην έρευνα και την καινοτομία. Τώρα συζητούμε για το φυσικό αέριο. Μιλάμε για αέριο, αλλά το αέριο είναι το φυσικό αέριο. Το υδρογόνο δεν είναι συμβατό ε, πολλές φορές με άλλες πηγές ενέργειας. Τώρα, αν συζητούμε για το υδρογόνο, το 95% ε, προέρχεται από φυσικό αέριο. Μόνο το 5% είναι από τις ανανεώσιμες. Η έρευνα λοιπόν στο υδρογόνο θα είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Επίσης, υπάρχει ανάγκη έρευνας και καινοτομία για την αποθήκευση των ε, ε, ανανεώσιμων. Θα πρέπει να έχουμε νέες επιλογές και για την αποθήκευση και για την ε, μεταφορά της ενέργειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, φυσικά είναι πολλές ερωτήσεις, οπότε σε ένα λεπτό είναι πολύ δύσκολο να απαντήσει κανείς ε, σε όλα τα θέματα, οπότε παρακαλούμε ε, σε ένα λεπτό να κάνετε την μεγαλύτερη, τη σημαντικότερη ερώτηση. Ο κύριος Ρόπε είναι ο επόμενος ομιλητής. Εδώ βρίσκομαι. Καλημέρα σας αγαπητή υποψήφια επίτροπε. Δίπλα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένας πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που κατασκευάζεται με, στη Λευκορωσία με ρωσικά κονδύλια. Παραβιάζει όλες τις διεθνείς συμφωνίες. Η Λευκορωσία αγνοεί τα stress test της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αποτελέσματά τους, διότι που διαπιστώνουν σοβαρά δομικά προβλήματα στο κατασκευή του εργοστασίου, τα οποία πρέπει να επιληθούν πριν ξεκινήσει να λειτουργεί το ηλεκτρικό αυτό, το πρινικό εργοστάσιο. Η Λευκορωσία δηλαδή θα προσπαθήσει να θέσει σε λειτουργία τον σταθμό αυτό, ενώ αυτός θα έχει προβλήματα. Τι βήματα θα λάβετε εσείς ε, ως ε, Επίτροπος ε, για να αποφύγουμε ένα νέο Τσερνομπίλ δίπλα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δικμές ασφαλείας στο Τσερνομπίλ έγιναν μετά από τη δυσλειτουργία των αντιδραστήρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρόμπα για την ερώτησή σας. Ξέρω ότι η κατασκευή αυτού του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ε, είναι ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα για όλους τους Λιθουανούς διότι βρίσκεται πολύ κοντά στην πρωτεύουσά σας. Και τι μπορούμε να κάνουμε με τα νέα πυρηνικά εργοστάσια που χτίζονται σε τρίτες χώρες μπορούμε να παράσχουμε βοήθεια ούτως ώστε η κατασκευή και η συντήρηση να γίνονται ε, βάσει των υψηλότερων προτύπων ασφαλείας. Επίσης μπορούμε να παρέχουμε οικονομική στήριξη σε εγκαταστάσεις τέτοιες τρίτων χωρών, ούτως ώστε οι διαδικασίες ε, που χρησιμοποιούνται εκεί να είναι ασφαλής. Και φυσικά μπορούμε να επιμείνουμε να πραγματοποιούνται όλα τα stress test και να λαμβάνονται σοβαρά τα αποτελέσματά τους. Ναι, θα λειτουργήσει αυτό το νέο πυρηνικό εργοστάσιο, αλλά εμείς θα παράξουμε καθοδήγηση για την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων ασφαλείας. Σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας, ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρασκευήσει υποστήριξη και στη Λιθουανία. Ούτω ώστε να είναι έτοιμη για πιθανές, ε, πιθανά περιστατικά εκτακτής ανάγκης. Ευχαριστώ. Uh, ε, up. Επερώτηση, κύριε Ρόπε. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Ήθελα μια πιο συγκεκριμένη απάντηση, αλλά αρκεί. Είναι γνωστό τη σπάση ότι το παρότι υποτίθεται ότι είναι μυστικό, ότι το ηλεκτρικό ρεύμα που θα παράγεται σε αυτό το εργοστάσιο στην ε, Λευκορωσία θα προορίζεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λουθονία βρίσκεται πολύ κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο αυτό και έχει δηλώσει ήδη ότι θα απαγορεύσει η εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύματο από αυτό το εργοστάσιο, διότι δεν πληρεί τα πρότυπα ασφαλεία. Τι θα γίνει με τα άλλα κράτη-μέλη, άλλε γειτονικέ χώρε και η δική σα, η Εστονία, η πατρίδα σα. Θα εισάγεται ή όχι αυτό το φθηνή ηλεκτρική ενέργεια θα αναλάβετε βήματα στο μέλλον, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαγορεύσει οριστικά ηλεκτρικό ρεύμα που δεν ε, προέρχεται από εγκαταστάσεις που πληρούν τα πρότυπα ασφαλεία. Ευχαριστώ. Κυρία Σίμψον. Ευχαριστώ κύριε Ρόμπεν. Ε, όπως ξέρετε η Εστονία, η Λετωνία και η Λιθουανία είναι σύμμαχοι στην ενεργειακή πολιτική. Έχω πολύ καλή συνεργασία με το δικό σας Υπουργό Ενέργειας και οι τρεις μας λοιπόν ανήκουμε στην περιοχή δίπλα ε, στη Λευκορωσία και συνεργαζόμαστε στενά ούτω ώστε να συγχρονίσουμε τις πολιτικές μας ε, και η διαδικασία συγχρονισμού θα είναι έτοιμη το 2025. Ε, είμαστε αισιόδοξοι. Ταυτόχρονα το πρόβλημα της διασυνοριακής ηλεκτρικής ενέργειας και του σχετικού εμπορίου δεν αφορά μόνο το πυρηνικά εργοστάσια, αλλά ε, δεν πληρώνουν τα τέλη για το διοξίδιο του άνθρακα και γι' αυτό έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πυρηνικά εργοστάσια, με τα ευρωπαϊκά εργοστάσια, συγγνώμη, τα εργοστάσια της Λευκορωσίας. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς επηρεάζεται ο ανταγωνισμό στι δικές μας αγορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπόρκια Ήτρε από το ID. Ευχαριστώ. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται για μια οικονομία βασισμένη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, όπως αναγνώρισε η υποψήφια επίτροπος, το φυσικό αέριο ε, παίζει ακόμα σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Ωστόσο, δεν υπάρχει σαφής κανονισμός όσον αφορά την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου. Κράτη-μέλη όπως η Ιαλία εξαρτώνται ακόμα από τις εισαγωγές ενέργειας όχι μόνο από τρίτες χώρες, αλλά και από άλλα κράτη-μέλη. Το υψηλό κόστος της εισαγόμενης ενέργειας επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της Ιταλίας ε, ε, των επιχειρήσεών της σε σχέση με τις επιχειρήσεις άλλων χωρών που μπορούν να βασιστούν σε χαμηλές ε, τιμές ενέργειας. Εσείς πώς σχεδιάζετε να διασφαλίσετε ότι οι εθνικές ενεργειακές πολιτικές για το φυσικό αέριο των κρατών μελών δεν θα παραβιάζουν τους κανόνες του ανταγωνισμού. Κυρία Σίμψον. Thank you for the question. There are European level um, agreements how we will um, Υπάρχουν ε, συμφωνίες ευρωπαϊκού επίπεδου για το άνοιγμα των αγορών μας ε, ε, διασυνοριακά. σε τέτοια περίπτωση η δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια μας λέει πώς θα μπορέσουμε να επιλύσουμε τους περιορισμούς των αγορών ε, στον τομέα της αγοράς ενέργειας. Ξέρω ότι σαφώς υπάρχει προσδοκία ορισμένα πράγματα που έχουν επιτευχθεί στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματο να αντιγραφούν και στην αγορά φυσικού αερίου και ειδικότερα η προσδοκία ότι και στην αγορά φυσικού αερίου θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τους καταναλωτές να έχουν δικαιώματα που έχουν ήδη οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό θεωρώ θα ήταν μια καλή ιδέα. Επερώτηση. Μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς ανθρακούχες εκπομπές ε, θα έχει κοινωνικο-οικονομικές ε, επιπτώσεις όχι μόνο σε κάποιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα δημιουργήσει συστήματα υποστήριξης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις χώρες που θα επηρεαστούν από τη μετάβαση ή θα περιοριστεί σε συγκεκριμένους κλάδους. Και επίσης αναφέρατε ότι οι υποδομές φυσικών αερίων θα πρέπει να συντηρούνται ανάλογα. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να σταματήσει χρηματοδότηση σε σχέση με ε, έργα υποδομών φυσικού αερίου ε, μέχρι τα τέλη του 2020, πώς την αξιολογείτε, θα είναι βιώσιμη η ευρωπαϊκή αγορά ακόμη και αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κυρία Σίμψον. Uh, τα έργα υποδομών θα είναι πολύ άριθμα. Αυτά που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνδέοντα στην Ευρώπη. Κάποια από αυτά θα χρειαστούν και συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ελπίζω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ε, υιοθετήσει μια δανειοδοτική πολιτική σύμφωνη με την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρωτήσατε τι μπορούμε να κάνουμε με τις κοινωνικές επιπτώσεις της μετάβασης. θα την στηρίξουμε. Και όταν αναφερόμαστε στο φυσικό αέριο, ε, σχεδόν ε, η μισή θέρμανση εξαρτάται από το φυσικό αέριο. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η ενεργειακή απόδοση είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο μείωσης του κόστους για τα νοικοκυριά μας. Ένας από τους κύριους λοιπόν επενδυτικούς στόχους θα είναι η ανακαίνιση των κτηρίων. όχι μόνο σε ορισμένες χώρες, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη και ειδικότερα για τις πολυκατοικίες, όπου θεωρούμε ότι οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και ε, κόστους είναι πολύ ψηλές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Στέγκρουντ. <clears throat> Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, κύριε Σίμψον, συγγνώμη, έχω κρυώσει, ελπίζω να με ακούτε. Εγώ είμαι νέα στο κοινοβούλιο, αλλά έχω έρθει από τον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα από την βιομηχανία της ενέργειας. Για πολλά χρόνια έχω εργαστεί με επενδύσεις, ενέργειες, αναλύσεις, συμπεριφορά καταναλωτών και ούτω καθεξής και ε, όταν διαβάζω τις ε, οδηγίες σας, ε, δηλαδή την εντολή σας ότι ο στόχος σας θα είναι να εξασφαλίσετε ότι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε προσιτή, αξιόπιστη και καθαρή ενέργεια, ναι, Πιστεύω πως όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με βάση προτεραιότητες και ναι, απαντήσατε ήδη σε κάποια από αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω διαφορετική ερώτηση. Εφόσον είμαι ως γυναίκα και προερχόμενη από την ενεργειακό τομέα, λέτε ότι το μερίδιο των γυναικών είναι 22% κατά μέσο όρο στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο και 32% στην ανανεώσιμη. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό και γιατί θεωρείτε πως είναι πρόβλημα. Κυρία Σίμψον. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Σύντομο σχόλιο Ε, λέτε πως ε, η καθαρή ενέργεια δεν είναι δυνατόν. Εγώ πιστεύω πως είναι, γιατί η ανανεώσιμη πηγή ενέργειας προέρχεται από τοπικούς πόρους, από τοπικές πηγές και ξέρω πως εκεί όπου ζω έχουμε πολύ προσιτή ε, ηλεκτρική ενέργεια από υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Είναι, είναι σαφώς ε, καθαρή, ασφαλής και προσιτή η ενέργεια αυτή. Βεβαίω θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια εκεί που υπάρχουν. Καλό παράδειγμα είναι ότι στο παραδοσιακό ενεργειακό τομέα Ε, η διαφορά είναι προφανής ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, αλλά στον τομέα της καθαρής ενέργειας και στην καινοτομία υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των δύο φύλων. Και αυτό είναι ένα από τα πρόσθετα ωφέλη της μετάβασης προς τις καθαρές πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ. αν ε, όλοι μπορούσαν να έχουν ε, πρόσβαση στην υδροελεκτρική ενέργεια, θα ήταν, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν ισχύει, δυστυχώς. Ε, ερώτησα γιατί θεωρείτε πως είναι πρόβλημα αυτό το ποσοστά και ποιο ποσοστό θα ήταν καλό εφόσον είμαστε στο 22% σήμερα ποιο θεωρείτε πως ήταν ένα δίκαιο νούμερο να φτάσουμε και πότε κυρία Σίμψον δεν ε, ε, έχουμε θέσει σχετικό στόχο, αλλά για όλους μας, εφόσον μιλάμε για μελλοντικά νούμερα, το σημαντικό είναι πόσες νέες θέσεις απασχόλησης θα δημιουργηθούν. για την ε, κλιματική με το, μετριασμό, τον, τι είδους θέσεις απασχόλησης θα είναι επίσης και από αυτή την άποψη πιστεύω ότι οι θέσεις στον τομέα της ενέργειας αλλά και στην έρευνα και στην κοινοτομία είναι το ίδιο κατάλληλες για τα δύο φύλλα. Η Ευρώπη πρέπει να μείνει σε ηγετική θέση στην πορεία προς την ουδετερότητα, κλιματική ουδετερότητα. Μάλιστα. Κύριο Σκέλη από το ΕΛΚ τώρα. Καλημέρα σας. Κυρία Σίμψον. Και ελπίζω και ελπίζω να ε, αισθάνεστε άνετα σε αυτή την καρέκλα που είστε μέσα προβολής και στα φώτα. Λοιπόν, ήμουν εισηγητής για τα ποσοστά ε, μέχρι το 2030. Ε, πώς ε, σκοπεύετε να φτάσετε στους στόχους. Είπατε ότι η Εστονία στοχεύει στο 42% μέχρι το 2030. Αυτό θα εντυπωσιάσει ακόμα και τους πράσινους. Ένας από τους στόχους νομοθεσίας ήταν η συμμετοχή των πολιτών ε, για μια μετάβαση ε, χωρίς διοξείδιο του άνθρακα. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβετε για να διευκολύνετε ε, τις νέες πρωτοβουλίες νοτόμες επιχειρήσεις αποκεντρωμένα και πώς θα κινητροδοτήσετε τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες σχετικά με την ίδια τους την κατανάλωση και τη συμπεριφορά να μεταβούν σε νέες ε, πηγές ενέργειας και να βοηθήσουν και συνολικότερα στην ενεργειακή μετάβαση. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Αυτό όντως ήταν ε, τμήμα του σχεδίου μας να συμμετέχουν περισσότερο οι πολίτες με τον τρόπο που εκείνοι θεωρούν σκόπιμο για να μειώσουν ε, την ενεργειακή τους κατανάλωση. Τώρα, ε, υπάρχουν υπολογιστές ε, ηλιακής ενέργειας που κοστίζουν πέντε φορές λιγότερο από ό,τι κάποια χρόνια πριν. Υπάρχει καινοτομία και στην Εστονία. Έχουμε εγκρίνει νομοθεσία που δίνει πρόσβαση στην αγορά τους πολύ μικρούς ε, παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόγραμμα λέγεται Plug and Play. Συνδέσου ε, στο δίκτυο και παίξε. Και έχουμε πολύ, πολλούς μικρούς παραγωγούς. Αυτό έγινε δυνατό διότι συζητήσαμε με τους διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην αρχή ανησυχούσαν, αλλά τώρα πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα. Η αγορά είναι πολύ ανοιχτή, ανταγωνιστική, ακριβώς γιατί έχουμε και ένα κόμβο δεδομένων, data hub, όπου συγκεντρώνονται όλοι οι παραγωγοί και οι καταναλωτές. τέτοιου είδους λοιπόν ε, πρωτοβουλίες βοηθούν πάρα πολύ τους πολύ μικρούς ε, παραγωγούς για να βγάζουν την ενέργεια που παράγουν στο δίκτυο. Και έτσι μας βοηθούν εμάς να πληρούμε τους στόχους που έχουμε για τις Μας Ευχαριστώ. Στην πραγματική ερώτηση ο κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σίμψον. Πολύ ενδιαφέρουσα η απάντησή σας μου φαίνεστε πάρα πολύ λογική και πάρα πολύ πρακτική. Ξέρετε ότι η μεγαλύτερη επίκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η γραφειοκρατία ε, και ε, το σχετικό άχθος. Πώς θα φροντίσετε στο δικό σας χαρτοφυλάκιο να μην προσθέσετε επιπλέον γραφειοκρατικό κόστος ε, που θα γονατίσει τις μικρομισές επιχειρήσεις και όσους ενδιαφερόμενους και αντιθέτως πώς θα τους βοηθήσετε για να ανθίσουν όλοι αυτοί οι φορείς. Νομίζω ότι το πακέτο για την καθαρή ενέργεια μας δίνει ένα πλαίσιο και τώρα καλούμαστε να εφαρμόσουμε τα εφιστάμενα μέσα και εργαλεία και να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτά δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους μικρούς παραγωγούς, ιδιώτες, να δίνουν την αγορά τους, ε, την ενέργεια μάλλον στην αγορά. Αυτό ισχύει και για άλλα στοιχεία. Για την ενεργειακή απόδοση, ας πούμε. Όπου απαιτεί όλα τα νέα κτίρια να είναι όχι απλώς αποδοτικά, αλλά να παράγουν και τα ίδια τα κτίρια ε, ένα κλάσμα της ενέργειας που θα καταναλώνουν στο μέλλον. Υπάρχουν τα κίνητρα και τα μέτρα, τώρα τα κράτη-μέλη καλούνται να τα εφαρμόσουν. Και να τα ανοίξουν για όλους τους ενδιαφερόμενους. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, next speaker is Mr. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Πεκαρίνεν από το Ρινιέν. Θα μιλήσω στα φιλανδικά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχηθώ ότι καλύτερο στην Επιτροπό. Πιστεύω ότι θα έχετε μεγάλη επιτυχία στη μελλοντική σας θέση. Τώρα τα σχέδια περί ενεργειακής ε, απόδοσης ε, μείωση εκπομπών του 40% είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέχρι το 2030 λέγεται. Ωστόσο, απέχει πολύ αυτό από το 50% ή το 55%. Πού πρέπει να εστιαστούμε στις μελλοντικές δράσεις. Στον τομέα ανταλλαγή εκπομπών, εμπορία εκπομπών ή στον κλάδο του καταμερισμού των βαρών. Μιλήσατε για τι ανανόσιμες πηγέ ενέργεια Ποια είναι η άποψή σα για τη βιοενέργεια που για μας τους Φιλανδούς είναι πολύ σημαντική μεταξύ των πηγαίνει μεταξύ των ανανεώσιμων. Ε, κυρία Σίμψον, ευχαριστώ κύριε Πεκαρινέν για την ερώτησή σας και θα σας απαντούσα και εγώ στα αισθανικά γιατί περίμενα να μου δοθεί δυνατότητα να χρησιμοποιήσω την μητρική μου γλώσσα. Αλλά όπως φαίνεται κανείς από την Εστονία δεν θα κάνει ερώτηση. Αλλά θα συνεχίσω αγγλικά για πιο εύκολα. Ρωτήσατε πώς θα επιτύχουμε ε, τη μείωση, τη, μεγαλύτερο, κατά μεγαλύτερο ποσοστό των εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου. Συμφωνώ ότι ο τομέας της ενέργειας ε, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί αυτή τη στιγμή το 75% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προέρχονται είτε από την παραγωγή είτε από την κατανάλωση ενέργειας. Αλλά υπάρχουν και άλλοι κλάδοι που θα πρέπει να συμβάλλουν. Το θέμα αυτό δηλαδή θα έχει πρώτη προτεραιότητα στην επόμενη Επιτροπή. Και στη δομή της νέας ε, θα υπάρχει ο εκτελεστικός ε, αντιπρόεδρος για το Green Deal, ε, ο κ. Τίμερμανς και θα συνεργάζονται μαζί του και άλλοι επιτροποί που θα ασχολούνται με την ενέργεια, τις μεταφορές, των περιβάλλον, τις γεωργικές υποθέσεις, την υγεία. Ε, ότι όλοι αυτοί θα ασχολούνται με αυτό το θέμα ε, δείχνει ότι είναι ο, κοινός μας στόχος. Ξέρω ότι ο αντιπρόεδρος Φρανς Τίμπερμανς ε, θα εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης του σημερινού συστήματος ETS. Σε το, υπάρχουν τομείς όπως οι οικοδομές, οι μεταφορές που δεν καλύπτονται ακόμα από αυτό το σύστημα, τα κτίρια και οι μεταφορές αλλά που θα μπορούσαν να συμβάλλουν. Κατά την άποψή μου, εγώ διακρίνω ωφέλη στην έξυπνη ενσωμάτωση, στην έξυπνη ολοκλήρωση. Ε, στενή συνεργασία δηλαδή μεταξύ πολλών κλάδων, με αποτέλεσμα χαμηλότερο ε, αποτύπωμα άνθρακα για το όπω οι μεταφορέ, ε, η βιομηχανία και φυσικά ο τομέας των κτηρίων, η ψήξη και η θέρμανση. Ευχαριστούμε. Επερώτηση. Ευχαριστώ. Η παγίδευση ε, άνθρακα ε, είχε σχετικές τεχνολογίες παγίδευσης άνθρακα δεν σημείωσαν την πρόοδο που αναμενόταν. Μία δυνατότητα ήταν η ε, απαλλαγή του άνθρακα από τα ορειτα δηλαδή από το διοξείδιο του άνθρακα παράγουμε συνθετικό προϊόν ε, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά έχοντας ε, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μπορούμε να μετατρέψουμε το διοξείδιο του άνθρακα σε μεθάνιο, το οποίο ε, μπορεί να αποτελέσει τρόπο αποθήκευσης του άνθρακα. Θέλετε εσείς να προωθήσετε αυτό τα τολμηρά έργα απαλλαγής από και εκπομπές. Ευχαριστώ κυρία Σίμψον. Ευχαριστώ κύριε Πεκαρίνεν. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι αναφέρατε αυτό το ζήτημα της ε, παγίδευσης και ε, αποθήκευσης και εκμετάλλευσης του άνθρακα. Διότι σίγουρα θα αποτελέσει ένα από τα θα αποτελέσει ένα από του μηχανισμού που θα μα βοηθήσουν να επιτύχουμε μέχρι το 2050 την ε, ουδετερότητα άνθρακα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιο έργο Ωστόσο υπάρχουν κάποια εμβληματικά έργα ανά τον κόσμο. Αυτό που ε, έχουμε εμεί ως πειραματικό έργο ε, είναι στο λιμάνι του Ρότερνταμ όπου προγραμματίζουν ε, υπεράκτια παγίδευση και αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Αν χρηματοδοτηθεί θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι το 2023. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε τέτοια έργα ακόμα, αυτό το Ρότερνταμ είναι το πιο κοντινό σε αυτή την τεχνολογία, ο λόγο που δεν υπάρχουν είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και οι αμφιβολίες που υπάρχουν όσον αφορά την αποθήκευση του άνθρακα. Και φυσικά η χρειαζόμαστε διαφορετικού στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Κοράου. Ανεξάρτητο. Με εγγεγραμμένος. Bene, lei Ευχαριστώ. Εσείς ως Επίτροπος Ενέργειας ε, θα έχετε ενώπιόν σας πολύ σημαντικές προκλήσεις. Ανάμεσα σε αυτές ήταν, ε, είναι ε, το θέμα των βιομηχανιών παραγωγής ενέργειας που παράγουν το 52% του διοξιδίου του άνθρακα. Και έχουμε επίσης την αναδιάρθρωση και των κτίριων που μέχρι τώρα γίνεται πολύ αργά και ανεπαρκώς υπαρχουν ε, ε, Υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία συνοδεύουν αυτές τις προκλήσεις. Πώς ε, σκοπεύετε να εντάξετε την κυκλική οικονομία στο θέμα της αναδιάρθρωσης των κτηρίων. Να σας πω και κάτι ακόμα για τις ενεργειακές κοινότητες που μου είναι πολύ προσφυλές σε θέμα. Μέσω της ιδιοποίησης της παραγωγής της ενέργειας οι, οι, καταναλωτές δεν είναι πια απλοί καταναλωτές, είναι και παραγωγή της ενέργειας με διάφορα πλονεκτήματα βέβαια. Πώς σκοπεύετε αυτά όλα να γίνουν δεκτά και να εφαρμοστούν και σωστά. Κυρία Σίμψον, διάφορες ερωτήσεις μου θέσατε και θα αρχίσω από την αρχή. Για την ε, ε, τηλεθέρμανση. Ναι, αυτό είναι μια από τα μεγαλύτερα, ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια τα οποία θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο να έχουμε περισσότερα πλέον εκτήματα από την τηλεθέρμανση. Μία από τις επιλογές είναι η αποτελεσματική συμπαραγωγή. Εάν μπορούμε να παράγουμε τόσο θέρμανση όσο και ηλεκτρισμό, τότε ήδη το 10% της ενεργειακής απόδοσης είναι ε, εφικτό. Επίσης, η βιοενέργεια για τη θέρμανση είναι επιλογή, η ευφυής ε, ε, επίσης ολοκλήρωση των τομέων για τη σύνδεση ε, των τομέων, καινοτομίες για τις αντλίες θέρμανσης κτλ. Όλα αυτά περιορίζουν το κόστος της θέρμανσης, αλλά το μεγαλύτερο μερίδιο είναι εάν όντως μπορέσουμε να ανακαινήσουμε τα κτίρια μας. 75% περίπου των ε, πολυκατοικιών, ε, δηλαδή των κτηρίων ε, με καταλήματα, είναι ανεπαρκή. Έχουν κατασκευαστεί τη δεκαετία του 80 και αν τα συγκρίνουμε με τα σημερινά, εκείνα τα παλιά χρησιμοποιούν, καταναλώνουν τη διπλάσια ενέργεια από ό,τι τα καινούρια. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι οι εξοικονομήσεις είναι ορατές, αλλά ταυτόχρονα μας λείπουν ε, χρήματα για την ανανέωση, για την ανακαίνιση και για την επιτάχυνση αυτής. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Καταρχά μπορούμε να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές γιατί σε κάποια κράτη-μέλη έχουν φεύρει ευφυεί τρόπους για να επελκύσουν ιδιωτικέ επενδύσεις και αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει και για τις υπόλοιπες χώρες. Ευχαριστώ. Επερώτησε κύριε Κοράου. Μάλιστα. Καταλαβαίνω πως ρώτησα πολλά πράγματα στην πρώτη ερώτηση και θα χρησιμοποιήσω και τη δεύτερη ε, επερώτηση για να εξειδικεύσω τις ερωτήσεις μου. Ε, για τις ενεργειακές κοινότητες, όταν μιλώ για εκδημοκρατισμό του ενεργειακού τομέα, αναφέρομαι στην ευκαιρία που έχουμε να χρησιμοποιήσουμε τους ε, πολίτες ως καταναλωτές και να μην τους θεωρήσουμε μόνο τη μετάβαση πώς, για τους μεγάλους παίκτες εσείς, πώς τους μεγάλους φορείς εσείς, πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη θέση για να προχωρήσετε προς αυτόν τον εκδημοκρατισμό της ενέργειας. Ναι, οι, κατα... μπορούν όντως να γίνουν ε, παραγωγή, μπορούν να παράγουν, να αποθηκεύουν και να πολλούν ενέργεια. Ε, και αυτό ε, σημαίνει ένα μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού που ζει σε πολυκατοικίες. Αυτή η μικροπαραγωγή λοιπόν, παραγωγή και κατανάλωση, είναι πολύ σημαντικό εκεί για να πετύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους. Είναι επίσης σημαντικό να δείξουμε ότι οι καταναλωτές μπορούν να ωφεληθούν από την μετάβαση και ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τις ε, πιο τελευταίες καινοτομίες. Ευρωπαϊκή καινοτομία όπως ας πούμε τα ηλιακά πλακάκια που παράγουν ε, και ε, ενέργεια. Ευχαριστώ κυρία Σίμψον. Σας ευχαριστώ για την αναφορά σας στη Γαλλικία στην αρχή Τη ομιλίας και τώρα θα συνεχίσω στα ισπανικά. Έχουμε το στόχο της διασύνθεσης του 15% για το 2030. Η διασύνδεση βελτιώνει τη μεταφορά των ανανεώσιμων από τη μια περιοχή στην άλλη. Αλλά στην Ευερική Χερσόνησο, για παράδειγμα, η διασύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη βρίσκεται μόλις στο 2,8%. Αν έχουμε λοιπόν ο στόχο το 15% και κάπου είμαστε στο 2,8%, ε, κάτι πάει στραβά είναι πολύ δύσκολο ο στόχος να καλυφθεί. Ε, ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα και χρονοδιαγράμματα που θα εγγυηθούν ότι θα καλύψουμε το 15% το 2030 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τι θα φέρετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. Και θέλω να σας ρωτήσω, ε, απαντήσατε πολλά για το φυσικό αέριο και κάποιες ερωτήσεις δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως επαρκώς. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι συμβατό με τις συμφωνίες του Παρισιού. Η κυρία Σίμψον. Ευχαριστώ κύριε Γκονσάλης Κασάρης. Πολύ σημαντικό το ερώτημά σας για τις διασυνδέσεις. ο στόχος του 10% αναβλήθηκε. Ήταν για το 2020 και στο μεταξύ για το 2030 αυξήσαμε το ποσοστό από 10% σε 15%. Τι μπορούμε να κάνουμε. Να προωθήσουμε την περιφερειακή συνεργασία και να χρηματοδοτήσουμε ε, την ε, κάλυψη αυτών των ε, κρίκων που λείπουν από την αλυσίδα η Ιβερική Χερσόνησος θα διασυνδεθεί από το Βυσκαϊκό κόλπο και αυτό χρηματοδοτείται από τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Αυτό δεν αρκεί, χρειάζεται περισσότερες συνδέσεις. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, διότι οι περιφέρειες αυτές που δεν είναι στο κέντρο γεωγραφικά της Ευρώπης χρειάζονται τέτοιου είδους συνδέσεις για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά αυτή η διασύνδεση από το βοσκαϊκό κόλπο νομίζω είναι μια πολύ καλή αρχή. Για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και κατά πόσο θα είναι χρήσιμο. Για το μακροπρόθεσμο στόχο μας της κλιματικής ουδετερότητας. Για την κλιματική ουδετερότητα θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο. Ε, στο υδρογόνο και σε αέρια που εκπέμπουν χαμηλό ε, ε, διοξίδιο του άνθρακα, όπως είναι και τα βιοαέρια. Και να δημιουργήσουμε και το δίκτυο. Πρέπει να ξέρουμε ότι μετά το 2030 όλα αυτά που θα φτιάχνουμε θα πρέπει να αντέχουν στο χρόνο Άρα σημαίνει ότι χρειάζεται μεγάλη έρευνα προς το υδρογόνο να διοικητευτεί. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Συνεχίζω με τις διασυνδέσεις και θα ήθελα να είμαι πιο συγκεκριμένος. Το είπατε κι εσείς η ίδια. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες για να καλύψουμε τους στόχους μας. Μιλήσατε αφηρημένα, αλλά υπάρχουν χώρες που δεν θα ποντάρουν ενδεχομένω σε αυτέ τι διασυνδέσεις. Η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει. Θα λάβει μέτρα για τα κράτη-μέλη που εμποδίζουν ε, να προχωρήσουν αυτέ οι διασυνδέσεις. Η κυρία Σίμψον. Φυσικά. Αυτή η στόχη για τις διασυνδέσεις ε, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι στόχοι δεσμεύουν όλα τα κράτη-μέλη όχι μόνο το 15% μέχρι το 2030, αλλά και άλλοι στόχοι. Για το ποιο τμήμα της διασύνδεσης και το εγώ εκεί θα είναι ανοιχτό στην αγορά. Και αν υπάρχει νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποχρεούνται όλα τα κράτη-μέλη να την εφαρμόζουν και να στοχεύουν στην κάλυψη αυτών των ποσοστών. Ευχαριστώ. Επόμενη μιλήτρια, κυρία Βάης. Να ευχαριστώ συγχαρητήρια για τον υποψηφιότητά σας και ευχαριστούμε για τις απαντήσεις. Είμαι εδώ ακριβώς μπροστά σας. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση για την αυξημένη ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Από όσο κατάλαβα από τη δική σας απάντηση στον κύριο Κέλλη, έχετε ήδη όλα τα εργαλεία και απλά αρκεί να τα χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη στην ε, επιστολή ε, αποστολή τη κυρία Βάντερ Λάιν μιλάτε για επιτάχυνση τη ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και οι κατευθυντήριε γραμμέ για την ενεργειακή απόδοση υιοθετήθηκαν πέρυσι και θα υλοποιηθούν σίγουρα. Επιβάλλουν διάφορε απαιτήσει ε, στα κτίρια για να επιτευχθεί ενεργειακή απόδοση στα κτίρια ε, μέχρι το 2021. Μέχρι το 2050 θα πρέπει όλα τα κτίρια να είναι ε, ουδέτερα από άποψη ανθρακά και ενεργειακά αποδοτικά. Ωστόσο έχουμε 1% ποσοστό ανακαινήσεων. Πώς θα επιταχύνεται ε, το ρυθμό αυτό για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των κτίριων. Θα ξανανοίξετε αυτή την οδηγία για υιοθέτηση ξανά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ κύριε Σίμψον. Ευχαριστώ. Το πρώτο εργαλείο που μπορώ να χρησιμοποιήσω ε, για την παρακολουθή της ενεργειακής απόδοσης ε, και του ρυθμού ανακαινήσεων είναι τα εθνικά σχέδια ενέργειας και κλίματος. Έτσι θα δούμε ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι για κάθε κράτος μέλος μέχρι τα τέλη του έτους. Ξέρω ότι υπάρχουν ανησυχίες ότι δεν θα καταφέρουν όλα τα κρατη να επιτύχουν τους στόχους. Αλλά έχουμε ακόμα τρει μήνες διαπραγμάτευση με τα κρατη ε, και παροχής ε, των βελτιστών συμβουλών. Φυσικά περιμένουν και συμβουλές από εμάς για το τι είδους ε, οικονομική στήριξη μπορούν να αναμένουν. Τέτοιου είδου δράσει μπορούμε εμεί να τι υποστηρίξουμε με διάφορου τρόπου από διάφορα ταμεία. Το μεγαλύτερο ταμείο για όλες τις ενεργειακές επενδύσεις θα είναι ο μηχανισμός συνδέοντας την Ευρώπη, το CEF. Ταυτόχρονα όμως ε, για τους αριθμούς ανακαινήσεις δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των κονδυλίων θα προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα. Θα πρέπει να υπάρξουν δάνεια υπό ευνοϊκούς όρους και φυσικά σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει νομοθεσία που θα επιτρέπει σε πολυκατοικίε να λάβουν τέτοια δάνεια, αν υπάρχουν ε, εκεί όπου υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτε. γιατί αυτέ οι πολυκατοικίε παρουσιάζουν συγκεκριμένε νομικέ δυσκολίε όσον αφορά την ε, λήψη δανείων. Οπότε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και διαθεσιμότητα δανείων. Επιπλέον των σχεδίων για τον άνθρακα. Ευχαριστώ. Επερώτηση, κυρία Βάη. Ναι, ευχαριστώ τα κτίρια με τη χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση συχνά κατοικούνται από ανθρώπους χαμηλών εισοδημάτων. Κάποια από αυτά τα κτίρια θα πρέπει να βγουν από να πάψουν να υπάρχουν. Πώς εσείς, τι θα κάνετε γι' αυτό, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι φτωχοί αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση σε ε, προσιτές, σε προσιτή κατοικία ε, και, ικανο, ε, και αξιοπρεπή. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Αυτός ο στόχος ανακαίνησης των αναποτελεσματικών κτηρίων, μη αποδοτικών κτηρίων αυτή τη στιγμή, ναι, πράγματι σε ορισμένα τέτοια κτίρια οι θερμοκρασίε το χειμώνα είναι κρύες γιατί είναι τόσο αναποτελεσματικά. Και σίγουρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους αυξημένους λογαριασμούς μετά από την ανακαίνωση. Ξέρω σε τέσσερα κράτη-μέλη υπάρχουν εθνικά σχέδια. επένδυση σε ανακαινήσεις ε, κοινωνικών κατοικιών. Διότι οι ένικοι είναι αυτοί οι οποίοι επηρεάζονται περισσότερο από τις υψηλές τιμές. Αυτή είναι μία από τις πρακτικές που μπορούμε να έχουμε υπόψη μας. Αυτό σημαίνει όμως ότι μετά από την ανακαίνιση θα μειώνεται το κόστος της θέρμανσης και θα επιτυγχάνονται ευκολότερα άνετες θερμοκρασίες. Ευχαριστώ. Next uh, speaker, uh, Rego. Επόμενη μιλήτρια, κυρία Ρέγκο, από την ΚΟΕ. Señora Σίμψον, Κυρία Σίμψον, εγώ ανησυχώ πολύ περισσότερο από ό,τι όταν έφτασα, κυρίως όσον αφορά την επίγουσα κατάσταση του κλίματος, το τι απαιτείται αυτό, απαιτείται λόγω αυτού και την ε, ρήξη και έλευθη αλλαγή ευρωπαϊκών πολιτικών που χρειάζεται. Ε, πριν από λίγο καιρό, ένα με μεγάλη ε, μια ομάδα μάλλον μεγάλων εταιριών μας επιβάλλουν ε, την πολιτική τους. Οι συνέπειες είναι σαφείς. Κλιματικές αλλαγές, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι υποφέρουν από την ενεργειακή φτώχεια και βεβαίως ε, πολιτικοί που έρχονται εδώ πέρα να υπερασπιστούν τα συμφέροντα αυτών των ε, μεγάλων εταιριών. Τα όσα εσείς μας προτείνετε δεν θα λύσουν την κλιματική αλλαγή. Ακόμα μια από τα ίδια μας προτείνεται Η πολυεθνική εθνικέ ενέργειε θέλουν απλά να σώσουν ε, τη δική τους, τις δικές τους επιχειρήσεις. Εσείς ε, ε, πρόκειται να κάνετε τίποτα ώστε να μετατρέψετε το ευρωπαϊκό μοντέλο σε μοντέλο βιώσιμο και που θα μπορεί να στηρίξει και τους πιο αδύναμους κοινωνία. Με ποια μέτρα ακριβώς θα το κάνετε αυτό. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας και πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η Επιτροπή είναι προσιλωμένη στην επίτευξη των κλιματικών στόχων και δεν είμαι εγώ μόνη που, ε, που είμαι υπεύθυνη για την ενέργεια. Πρόκειται για τη δέσμευση της υποψήφιας Προέδρου, πρόκειται για γενικούς και στόχους και για μια ε, γενική προτεραιότητα που είναι η κύρια ευθύνη του Αντιπροέδρου Φραντ Τίμερμανς που είναι υπεύθυνο για αυτά τα θέματα. Και θα υπάρξει κλιματική νομοθεσία και σαφές πρόγραμμα δράσης. Η δική μου ευθύνη ως Επιτρόπου για την Ενέργεια είναι να εξασφαλίσω ότι η ότι, θα, ότι ότι θα επιτύχουμε μάλλον όλους αυτούς τους στόχους και την ενεργειακή απόδοση ότι θα έχουμε ε, προσιτέ τιμέ και ότι η βιομηχανία μα θα είναι ανταγωνιστική σε σχέση με άλλε περιοχέ του κόσμου. Και βεβαίω, μία από τι δικέ μου αρμοδιότητε θα είναι το να μπορώ να έχω επαφή μέσω του ενεργειακού διαλόγου. Γιατί πρέπει έτσι να δώσουμε κίνητρα και στου εταίρου μα, δηλαδή να κάνουν και εκείνοι τα αντίστοιχα και να μπορέσουμε έτσι με αυτά τα εργαλεία να συνεργαστώ δηλαδή στενά με τα κρατημέλη και να τα παροτρύνω να, να υψώσουν τον πύχη, να βάλουν ψηλότερους στόχους, να συνεργαστώ με τους ε, συναδέλφους επιτρόπους και να εξηγήσω τη μεγαλύτερη έλλειψη χρηματοδότησης αυτή τη στιγμή αφορά την ενεργειακή απόδοση, ότι θα πρέπει να υπάρξει αύξηση όμως της χρηματοδότησης και για την έρευνα και την ανάπτυξη. Σε αυτά ε, δεσμεύομαι. Αλλά ο γενικός μας και στόχος είναι μέχρι το 2050 η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι η Ευρωπαϊκή Ήπειρος να είναι η πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος. Ευχαριστώ. Επερώτηση. Φαίνεται να υπάρχει μια μικρή αντίφαση στα όσα μας λέτε. Θα είμαι πιο σαφής και πιο ευθύς. Αυτό που είναι απλό, υπάρχει άμεση συσχέτιση ανάμεσα στην ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές. Και η ενέργεια είναι στα λίγα χέρια που έχουν εκμεταλλευτεί από την εξωτερήκευση του περιβαλλοντικού κόστους και των ενεργειακών πολιτικών της Ένωσης για να κάνουν business και μας άφησαν ε, εκπομπές που έχουν συμβάλει στο να είμαστε αυτή τη στιγμή σε ε, ε, ακραίο κίνδυνο ολόκληρος ο πλανήτης τι θα κάνετε εσείς για όσον αφορά την αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου, δηλαδή απόδοση, δημοκρατικός έλεγχος και μείωση της παραγωγής και της κατανάλωσης. Εσείς από με ποια μεριά είστε, με τη μεριά του Ένι, με τρόλα, τη, της Γκαστέρα, της Waterfall και όλων των άλλων ομίλων ή με την πλευρά των όσων αγωνιζόμαστε για ένα ζωντανό πλανήτη για τις επόμενες γενιές. Thank you. Well, energy consumers will be heart of our... Um, um, Η κατανάλωση ενέργειας είναι στην καρδιά της ενεργειακής πολιτικής και αυτό είναι το έργο μου. Το να μπορέσουμε να έχουμε προσιτή ενέργεια και αυτό μέσω της διαφοροποίησης των πηγών. με την πολιτική διασύνδεση των ενεργειακών ε, δικτύων, την ισορροπία της ε, παραγωγής και βέβαια και τις επενδύσεις ε, που θα βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις συνδέσεις του, εκεί όπου δεν υπάρχουν, να τις δημιουργήσουμε έτσι ώστε όλοι να ωφεληθούμε εφόσον υπάρχει ε, στην νότερη συνεργασία, καταρχάς σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά και στη συνέχεια και από την εσωτερική αγορά, που θα ε, προσφέρει πιο ανταγωνιστικές τιμές στους καταναλωτές. Μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας μόνο όταν υπάρχει ε, δημόσια αποδοχή και στήριξη. Αυτό θα υπάρξει από τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι θα δουν πως όλα αυτά οδηγούν σε ανταγωνιστικές τιμές. Κυρία Γκρίφιν, Ευχαριστώ. Στην περασμένη θητεία καταπολέμηση της ενεργειακής στόχιας για πρώτη φορά κατοχυρώθηκε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περίπου 50 εκατομμύρια ευρωπαϊκά νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματο. Και το 2019 χρειάστηκε να διαλέξουν αν θα φάνε, ε, αν θα θερμάνουν ή αν θα ψήξουν τα σπίτια τους. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που πεθαίνουν από τη ζέστη γιατί δεν έχουν λεφτά να ανάψουν το ε, κλιματισμό. Υπάρχουν ε, σχέδια που έχουν υποβάλει τα κρατημέλη, αλλά είναι ανεπαρκή. Πώς ε, προτίθεστε να βελτιώσετε αυτή την κατάσταση και τι μέτρα θα προτείνετε για να συμμετέχουν ουσιαστικά οι ενδιαφερόμενοι. Ποια είναι η τεχνική υποστήριξη που θα προτείνετε για την ανταλλαγή καλών πρακτικών από χώρα σε χώρα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ε, θα έχουμε τα υψηλότυπα πρότυπα στην φιλοδοξία μας και στην καρδιά κάθε ενεργειακής πολιτικής θα είναι οι άνθρωποι, οι πολίτες και κυρίως ε, αυτοί που είναι στην ενεργειακή φτώχεια. Η κυρία Σίμψον. Σας ευχαριστώ. Μπορώ να σας διαβεβαίωσω ότι η έκθεση που κάνατε στην προηγούμενη θητεία έθεσε ένα πολύ καλό παράδειγμα για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες. Αυτό θα είναι και τμήμα των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα. Λαμβάνουμε υπόψη και ε, εκείνου που πλήττονται από την ενεργειακή φτώχεια και δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν το ρεύμα ή τη θέρμανση. Αυτό το καιρό τα σχέδια είναι στο αρχικό στάδιο. Θα δούμε τα τελικά πώς θα οριστικοποιηθούν στα τέλη του έτους. Και αυτό θα είναι και τμήμα των ετησίων εκθέσεων επίσης. Υπάρχει και η ε, κατάσταση όπου κάθε κράτος μέλος ορίζει την ενεργειακή φτώχεια με διαφορετικό τρόπο. Και θα πρέπει και εκεί ε, το παρατηρητήριο για την ενεργειακή φτώχεια να μας δώσει μια συγκεκριμένη ε, πρόταση, ένα συγκεκριμένο ορισμό για το πώς θα καλύψουμε αυτό το θέμα ενιαία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μια συμπληρωματική ερώτηση. κυρία Γκρίφιν, ευχαριστώ. Χαίρομαι που επιτέλους θα έχουμε και έναν ορισμό για την ενεργειακή φτώχεια. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω εσείς πώς ε, σκέφτεστε να βελτιώσετε αυτά τα προσχέδια. Γιατί ε, είναι ευρύ το φάσμα. Ορισμένα είναι πολύ ικανοποιητικά, πολύ επαρκή και κάποια άλλα τελείως ανεπαρκή. Ποια είναι η τεχνική βοήθεια που δίνεται και ποια κίνητρα και μια πολιτική ερώτηση έχω να σας κάνω. Γιατί πιστεύω ότι η ενέργεια δεν είναι απλώς ένα εμπόρευμα. Είναι ένα βασικό κοινωνικό δικαίωμα. Ως υποψήφια επίτροπος για την ενέργεια για 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, εσείς τι πιστεύετε ότι είναι η ενέργεια. Ευχαριστώ. Κυρία Σίμψον. Συμφωνώ ότι η ενέργεια ε, μας εντάσσει στην κοινωνία και καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι μια υπηρεσία πάρα πολύ απαραίτητη. Ταυτόχρονα, όταν μιλάμε για ενεργειακή φτώχεια, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ενέργεια ως ε, εμπόρευμα. Υπάρχουν και άλλα στο τιμολόγιο. Είναι τέλη, είναι φόροι, είναι ε, συμμετοχή για ε, τα δίκτυα. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε ακριβώς για αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό της θέρμανσης. Μπορούμε να βρούμε πιο αποτελεσματικούς τρόπους θέρμανσης. Δεν μπορεί να γίνει παντού, ούτε από τη μια μέρα στην άλλη. Υπάρχουν όμως διαφορετικές τεχνολογίες που μειώνουν το κόστος της θέρμανσης. Και φυσικά με τις ανακαινήσεις των κτηρίων θα έχουμε σημαντική πρόοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Παρούς από τους Πράσινους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Σίμψον που βρίσκεστε εδώ σήμερα μαζί μας. Θα συνεχίσω στα γερμανικά. Έχουμε διαπιστώσει ότι προ ένα κόσμο μηδενικών εκπομπών και με ανανεώσιμε ε, πηγέ ενέργεια χρειαζόμαστε περισσότερο φυσικό αέριο από ποτέ. Οπότε χαίρομαι που στι γραπτέ απαντήσει συμπεριλάβατε το Energy Efficiency First ω αρχή ε, που θα ισχύει για την υποδομή. Συμφωνώ για τις υποδομές. Και τώρα μια συγκεκριμένη ερώτηση. Λιγότερη, συγγνώμη. Ε, εσείς ε, μπορείτε να μας πείτε θα διασφαλίσετε ότι οι επενδύσεις μέσω ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή για τα έργα κοινού συμφέροντος είναι σαφές ότι θα ε, κατευθύνονται θα, από την αρχή Energy Efficiency First ε, τι θα γίνει με, τα εκτός χρήσης, ε, με τις εκτός χρήσης εγκαταστάσεις ε, που είναι απερχαιωμένες ε, για να πάμε σε ένα νέο κόσμο. Θα θέλουμε να μας αξιολογήσετε αυτό το πώς θα εφαρμόζεται η αρχή Energy Efficiency First. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Um, για τις επενδύσεις που θα προέλθουν από διάφορες πηγές και η μία πηγή θα είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το μέρος της που θα ονομαστεί η Κλιματική Τράπεζα στο μέλλον. Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τους κλιματικούς μας στόχους. Είναι σαφές ότι για να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα η προτεραιότητα θα είναι προτεραιότητα θα έχουν τα έργα που επενδύουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ενεργειακή απόδοση και στα δίκτυα. Για να επιτύχουμε λοιπόν τους στόχους μας χρειαζόμαστε καλύτερες συνδέσεις. Γι' αυτό το λόγο οι επενδύσεις ε, στα δίκτυα θα καταστούν απαραίτητες. Τώρα για τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΣΕΦ. Παρατηρούμε ότι σε σύγκριση με πριν από περίπου δύο χρόνια παλιότερα, το φυσικό αέριο, τα έργα φυσικού αερίου θα είναι όλο και λιγότερα. Και ενώ θα πολλαπλασιάζονται τα έργα ανανεωσιμών πηγών ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή είναι η τάση αυτή τη στιγμή που διακρίνουμε σαφώς. Και πιστεύω ότι ε, στην τρέχουσα επιτροπή, στη θητεία της τρέχουσας επιτροπής, θα έχουμε έναν τέταρτο γύρο PCI και περισσότερα έργα σε σχέση με την προηγούμενη. Ευχαριστώ. Ε, Επερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Αναφερθήκατε στην κλιματική τράπεζα μόλις και τους, ε, στους κλιματικούς μας στόχους. Έχω μια ερώτηση. Η στρατηγική για το μεθάνιο, ε, το μεθάνιο σήμερα είναι σημαντικό κομμάτι, όπως εκτιμάτε, για 15 έως 20% ε, το, διότι το μεθάνιο είναι υπεύθυνο για την υπερθέρμανση, ε, παραμένει περισσότερο στην ατμόσφαιρα από ό,τι παλιότερα. Αλλά παρέχει παρόμοιε δυνατότητε με το, με το φυσικό αέριο. Λένε όμως ότι χρειαζόμαστε διαφοροποίηση, αλλά ε, τερματικά διαφοροποίηση των παρόχων. Ποια είναι η στρατηγική για να παρεμποδίσουμε να, να μην υπονομεύσουμε τους κλιματικούς μας ε, στόχους χρησιμοποιώντας το μεθάνιο. Ευχαριστώ. Κυρία Σίμψον. Πράγματι, η διαρροή μεθανίου είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε εδώ στην Ευρώπη. Είμαστε σε χειρότερη θέση σε σύγκριση με τους κυρίους εταίρους μας. Μπορούμε να μάθουμε από τις εμπειρίες τους. Θα υπάρξουν πρωτοβουλίες στον τομέα του μεθανίου και στη διαρροή του μεθανίου. τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εμπλακούν στενά σε αυτή τη στρατηγική. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ. Η κυρία Τσέχ από την ομάδα Renew Europe. Σας ευχαριστώ η εκλεγμένη πρόεδρος ε, Φόντερ Λάιν είπε ότι η πολιτική θέλει να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει πολιτικό χαρακτήρα και γεωπολιτικό. Το ενεργειακό προφίλ είναι πολύ σημαντικό και η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν είναι ενωμένα τα κράτη-μέλη, όταν θέλουν να κάνουν επίσης την Ευρώπη πιο πράσινη, αλλά θα πρέπει όλα αυτά να φαίνονται και στα σχέδια των κρατών μελών που δεν επαρκή παρόλο που υπάρχουν κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις. Ορισμένα κράτη-μέλη φοβούνται ε, τον κίνδυνο και υπάρχει κίνδυνος να ενταθεί το χάσμα ε, Ανατολής Δύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με χαρά άκουσα ότι η Εστονία υποστήριξε ε, το στόχο για την ουδετερότητα και ρωτώ ως Επίτροπος ποια είναι τα μέτρα που θεωρείτε απαραίτητα για να ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη που έχουν μείνει πίσω στις δεσμεύσει τους να αναθεωρήσουν τους εθνικούς στόχους ε, ε, γενικότερα. Η κυρία Σίμψον. Ε, ευχαριστώ. Καταλήν ε, για όλα αυτά τα καλά νέα που μας είπες ότι έμαθες τώρα για την Εστονία. Εγώ δεν έχω ίντερνετ εδώ και δεν το ήξερα. Και αυτό είναι η απάντηση σε προηγούμενες ερωτήσεις. Και χαίρομαι γι' αυτό. για τα εθνικά ε, σχέδια ενέργειας και κλίματος, αυτά τα NECP. Βλέπουμε ότι τα διάφορα κράτη-μέλη δεσμεύονται σε διάφορα επίπεδα. Και αυτό γιατί η αφετηρία, όπως είπαμε, είναι διαφορετική από την οποία ξεκινάει το κάθε κράτος. Και τα κράτη έχουν διαφορετικό ενεργειακό μείγμα. Ε, κάποια εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα. Και είναι κλάδος της τοπικής τους, τους βιομηχανίας. αλλά και του κοινωνικού ιστού. Υπάρχουν συστήματα, ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης κτλ. Ε, και χρειάζονται ειδική βοήθεια. Θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Καθώς πλησιάζει το τέλος της ακρόασης, θα ήθελα και πάλι να επαναφέρω το θέμα και να αναφέρω ε, το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης. Ε, ρώτησαν πολύ γιατί δημιουργήθηκε και είναι ακριβώς ένα νέο μέσο και εργαλείο που βοηθάει εκείνες τις χώρες μέλη που έχουν πρόβλημα και έχουν και περιοχές ε, που παράγουν άνθρακα για να προετοιμαστούν να καταλήψουν τα στερεά ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι διαφορετικό από το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης που έρχεται να βοηθήσει εφόσον έχουν χαθεί οι θέσεις εργασίας. Το συγκεκριμένο Ταμείο ε, θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να χαράξουν τη σωστή στρατηγική και θα αποτελέσει και ένα γερό εργαλείο στη διαπραγμάτευση για τους στόχους με τα κράτη-μέλη. Και το επόμενο τρίμηνο ε, συνεχίζονται ακόμα οι διαπραγματεύσεις. Και στόχος είναι να έχουμε όσο γίνεται πιο φιλόδοξους στόχους ακριβώς. Ευχαριστώ. Um, Συμπληρωματική ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό να κινητροδοτήσετε τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα εκείνα που έχουν φτωχέ περιφέρειες, να αναθεωρήσουν την ενεργειακή πολιτική για να διευκολυνθεί η μετάβαση. Και περιμένω εδώ τις προτάσεις σας. Επίσης, θα ήθελα να δώσω συνέχεια σε κάποιες ερωτήσεις προηγουμένων συναδέλφων για τη μείωση εκπομπών ε, στις κατοικίες και στις μεταφορές στις χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης οι υποδομές μεταφορών και κατοικίες ε, παράγουν ε, πολλούς ρήπους σε σχέση με άλλες περιφέρειες. Θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία με την κυρία Φερέιρα και άλλους επιτρόπους. Η κυρία Φερέιρα έχει την περιφερειακή ανάπτυξη, ε, καθώς επίσης και το μελλοντικό ή τη μελλοντική επίτροπο για τις μεταφορές. Πώς σκέφτεστε να συνεργαστείτε ε, και ποια είναι τα σχέδιά σας ε, για τη μελλοντική σας αυτή συνεργασία. Η κυρία Σίμψον. Ευχαριστώ. Εγώ θεωρώ ότι δουλεύω πάρα πολύ καλά ομαδικά και προσβλέπω ε, στη συνεργασία όχι μόνο με τους συναδέλφους επιτροπούς αλλά και με το κοινοβούλιο σας και με τα κράτη-μέλη γιατί χωρίς αυτή τη συνεργασία δεν πρόκειται να φτάσουμε σε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους. Στην προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπος Άριας Κανιέτε ήταν αρμόδιος και για το κλίμα και για την ενέργεια. Ε, στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστώ στενά με τον εκτελεστικό ε, αντιπρόεδρο κύριο Τίμερμανς που είναι αρμόδιος για την Γενική Διεύθυνση Κλίματος. Ο κύριος Κανιέτε ήταν αρμόδιος για δύο γενικές διευθύνσεις, ενέργεια και κλίμα βλέπω χώρο για ευφύ ολοκλήρωση σε τομεί όπω είναι οι μεταφορές, η στέγαση, η θέρμανση, η ψήξη των κτίριων, αλλά και στη βιομηχανία. Και αυτή είναι και η μελλοντική δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η φιλοσοφία να συνεργαζόμαστε σε διαφορούς τομείς ε, και έτσι διακλαδικά. Ευχαριστώ. Thank you too. Now, uh, last speaker. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ομιλητής ε, για σήμερα. Η κυρία Σπυράκη από το ΕΛΚ. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Επίτροπε, είμαι εδώ. Επειδή είμαι η τελευταία που ζήτησα το λόγο, θα ήθελα να επιμείνω σε δύο θέματα που σχετίζονται με τον κοινό μας στόχο για τον άνθρακα, για την ουδετερότητα. Πρώτα απ' όλα, το Ταμείο Μετάβασης, Δίκαιης Μετάβασης, πότε θα δημιουργηθεί, τι πρικοδότηση θα έχει και πώ οι ε, 41 περιφέρειε τη Ευρώπη που εξαρτώνται από τον άνθρακα θα επιφοληθούν από αυτό. Η δεύτερη σχετική ερώτηση, σύμφωνα με την ε, πρόεδρο Ursula von der Leyen, τα σχέδια τη Κομισιόν για τη δημιουργία ε, ενός φόρου άνθρακα που έχει σκοπό τη μείωση της διαρροής άνθρακα στα σύνορα ε, και να βελτιώσει την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Μπορείτε να μα δώσετε περισσότερε λεπτομέρειε για αυτό το θέμα επίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Σίμψον. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ε, Μιλήσατε για το Ταμείο Δίκαιη μετάβαση πρώτα απ' όλα. Αυτό το Ταμείο αναφέρθηκε και στη δική μου επιστολή αποστολής. Ο Επίτροπος που θα υλοποιήσει και θα προωθήσει το σχέδιο θα είναι η Επίτροπος Φεραίρα. Εγώ θεωρώ ότι το Ταμείο Δίκαιες Μεταβάσεις θα επικεντρωθεί στο έργο για τις βασικές περιοχές, για τη μετάβασή του. Θα βοηθήσει και τα μικρά νησιά που δεν έχουν σύνδεση με την υπηρετική Ευρώπη. Έτσι θα βοηθηθεί κάθε περιοχή να εξοπλιστεί, να προετοιμαστεί καλύτερα για τη μετάβαση. Από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανόσιμες πηγές ενέργειας. το ακριβές ποσό που θα έχει αυτό το ταμείο είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση, αλλά επειδή θα ενταχθεί στο επόμενο πολιτισμο δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι μια πρωτοβούλια που θα συζητήσουμε τις πρώτες ήδη εβδομάδε από την, τις θητείες της επόμενης Κομισιόν. Προβλέπω λοιπόν ότι μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα έχουμε ήδη ε, συγκεκριμένες απαντήσεις. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ ώστε να προκοδοτηθεί επαρκώ, ώστε να υποστηρίξει αυτές τις περιοχές για να προετοιμαστούν ε, για τη μετάβαση. Για την, ε, τον συνοριακό φόρο άνθρακα ε, είναι συνεργατικό το έργο αυτό. Απαιτείται συνεργασία πολλών επιτρόπων, εμπορίου, οικονομικών και θα συμβάλλω και εγώ φυσικά. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας αναλύσω περισσότερο. Κυρία Σπυράκη, επερώτηση. Λοιπόν, σα υποβάλλω μια ερώτηση γιατί θέλω να μου δώσετε λεπτομέρειε όσον αφορά την υλοποίηση και τη λειτουργία του επωνομαζόμενου μηχανισμού, ε, του συνοριακού μηχανισμού. Γιατί ξέρω ότι η, υποψήφια επίτροπο ε, δεν μπορούσε να απαντήσει στην ερώτηση. Υπάρχει κάποιο είδου προετοιμασία σε αυτή την ε, επιτροπή για να αρχίσουμε ε, την, ε, τις εργασίες ή απλά είναι ένα θέμα που αναφέρεται. Ευχαριστώ. Ο συνοριακός φόρος για τον άνθρακα ως θέμα πρέπει να αντικαταστήσει το σημερινό μηχανισμό ε, και να είναι καλύτερος από αυτό το σημερινό μηχανισμό που ασχολείται με τη διαρροή άνθρακα. Δεν υπάρχει κάποιο οριστικό σχέδιο Υπάρχουν πολλές ιδέες. Ακούμε και απόψε από διάφορα κράτη-μέλη που έχουν συγκεκριμένα προβλήματα αθέμη ανταγωνισμού. Αλλά αυτός ο συνοριακός φόρος ε, άνθρακα θα πρέπει να είναι συμβατός με τους κανόνες του ΠΟΕ. Δεν πρέπει να περιορίζει το διεθνές εμπόριο. Ξέρω ότι αυτός ο συνεργός φόρος άνθρακα μπορεί να εξεταστεί και ανακλάδο και περιφερειακά. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου κλείνουμε τα δικά μας εργοστάσια και ξαφνικά εισάγουμε ε, ενέργεια που παράγεται με άνθρακα από άλλες χώρες όπως ε, στον τομέα του ηλεκτρικού ρεύματος. Ε, μιλάμε για περιφερειακές, τοπικές αγορές. Έχουμε μια τέτοια υπόθεση του ανταγωνισμού ουσιαστικά, όπως συμβαίνει με την Ισπανία και το Μαρόκο. Αυτές είναι οι τομεακές υποθέσεις που πρέπει να διαπραγματευτούμε και να αναλύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται ο γύρος ερωτήσεων. Κυρία Σίμψον, έχετε πέντε λεπτά για, τις τελικές σας, για την τελική σας παρουσίαση. Οπότε είστε έτοιμοι, έχετε τον λόγο. Είμαι έτοιμη. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, καλημέρα και στους Ευρωπαίους που μας βλέπουν από το διαδίκτυο. Ευχαριστώ για αυτή την πολύ σημαντική ακρόαση, τουλάχιστον για μένα. Ήταν ε, πολλές ερωτήσεις. Ελπίζω να κατάφερα να απαντήσω καθαρά στις ερωτήσεις σας. Ελπίζω να κατάφερα να εκφράσω και να διατυπώσω καθαρά τι ανησυχίε μου. Εγώ πιστεύω ακράδαντα στη συνεργασία μεταξύ επιτρόπων και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο σημερινός διάλογος ε, θεωρώ ότι δεν σταματά εδώ, δεν είναι παρά μια αφετηρία για μια ισχυρότερη, ε, μόνιμη συνεργασία εφόσον ε, διοριστώ ως Επίτροπος και προσβλέπω στη συνεργασία μας, στις συναντήσεις μεταξύ μας ως βασικό κομμάτι της δουλειάς μου. Απόλαυσα πολύ τις συζητήσεις μας κατά την Προεδρία της Εστονίας ε, το 2017. Είχα στα χέρια μου το, ως ε, Επίτροπος για ε, ενός χορτοφυλακίου που περιλαμβάνει μεγάλο κομμάτι ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Θα φροντίζω να ενημερώνεστε, να παίρνουμε τη γνώμη σας και να συμμετέχετε Σήμερα επιβεβαιώνεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα είναι μεγάλο σύμμαχο για την πρόθεση του Green Deal που θα διαμορφώσει το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσατε τι ιδέε, του στόχου μου για το μέλλον στην εναρκτήρια μου, μου δηλώσει και μεταξύ των απαντήσεών μου σε ερωτήσει σα θα ήθελα να τονίσω ορισμένα σημεία. Είναι σαφές ότι η βασική ανησυχία είναι το κλίμα. Ε, μεταξύ σας. Αν δεν λάβουμε συγκεκριμένα βήματα τώρα, το μέλλον θα είναι σκοτεινό. Πρέπει να δράσουμε τώρα. Γι' αυτό το λόγο η νέα πρόεδρος έχει προσδιορίσει το European Green Deal ως βασική προτεραιότητα. Πρώτη προτεραιότητα της επόμενης Επιτροπής. Θεωρώ ότι είναι σαφές ότι η ενεργειακή πολιτική θα βοηθήσει κέρια στην εκπλήρωση αυτών των προτεραιοτήτων και αφού το 72% των εκπομπών οφείλονται στην ενέργεια, η Ενεργειακή Ένωση θα παραμείνει ένα σοβαρό θεμέλιο για την Πράσινη Συμφωνία, διασφαλίζοντας ότι θα επιτευχθούν οι φιλοδοξίες ε, σε επαρκέ επίπεδο μέχρι το 2030 και πέραν αυτού. Η αποτελεσματική υλοποίηση τη υπάρξη νομοθεσία, ειδικότερα του πακέτου καθαρή ενέργεια, θα είναι η βασική οδό ε, για να αυξήσουμε τι φιλοδοξίε. Επίση, θα ήθελα να τονίσω ότι θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε κάποια ισορροπία για την ολοκλήρωση της, ε, ε, Ευρωπαϊκής, της Ενεργειακής Ένωσης και όλων των διαστάσεών της. Η Ενεργειακή Ένωση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για βιώσιμη, αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια για τους πολίτες μας. Έχει δημιουργήσει ένα μοναδικό νομοθετικό πλαίσιο ενέργειας και κλιματικής διακυβέρνησης πάνω στο οποίο θα πρέπει να χτίσουμε τις μελλοντικέ μας δράσεις. Οι μελλοντικέ μας δράσεις θα εστιαστούν στην ενεργειακή απόδοση, την πρώτη αρχή, και στην επιτάχυνση της ε, καθαρής ενέργειας της εφαρμογής της σε όλες τις οικονομίες. Θα βασίσουμε το σύστημα παραγωγής ενέργειας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην έξυπνη ολοκλήρωση ε, ηλεκτρικού ρεύματος ε, μεταφορών και κτηρίων. Η εσωτερική αγορά θα βασιστεί σε συνεργασία και η διεθνής διάσταση είναι σημαντική για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Στονίσατε επίση, πόσο σημαντικέ είναι οι τεχνολογικέ πρόοδοι και εγώ θα εστιαστώ σε αυτό. Είναι αδιανόητο η μετάβαση να βασιστεί μόνο σε κανόνε και σε ρυθμιστικά πλαίσια. Η Ευρώπη θα γίνει κλιματικά οδέτερη μέχρι το 2050 και μέσω τη καινοτομία, τη έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Με αυτόν τον τρόπο επίση θα ενισχύσουμε και τι βιομηχανικέ μα δυνατότητε. Πολλοί από εσά αναφέρατε ε, την καταπολέμηση τη αδικία ε, στον τομέα τη ενέργεια και τη ένδυα στον τομέα τη ενέργεια. Δεν μπορούμε να δεχθούμε εκατομμύρια Ευρωπαίοι να μην μπορούν να πληρώσουν του λογαριασμού του ή να βλέπουν να φουσκώνουν οι λογαριασμοί του. Είναι θέμα αλληλεγγύη. Και έτσι διασφαλίζεται και η δημόσια στήριξη που χρειαζόμαστε για τη μετάβαση. Οποιοδήποτε βήμα θα κάνουμε από εδώ και πέρα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τον καταναλωτή. Χρειαζόμαστε την υποστήριξή του, την κατανόησή του. Πολλοί από εσά επίση ρωτήσατε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για συγκεκριμένε περιφερειακέ ή εθνικέ καταστάσει. ειδικότερα για τι πιο ευάλωτε περιοχέ και τι μικρότερε χώρε. Μαζί είμαστε ισχυρότεροι. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για ένα καλύτερο μέλλον. Κανένα κράτο μέλο δεν πρέπει να μείνει πίσω καμία περιφέρεια. Γι' αυτό εγώ θα προσπαθήσω να υλοποιηθεί το Ταμείο Δίκαιης μετάβαση, ώστε να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μέχρι στιγμή μίλησα στα αγγλικά, αλλά θα ήθελα να κλείσω στη μητρική μου γλώσσα, στα εστονικά. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ, σε εποχές που η Ευρώπη μεταβάλλεται. Ε, σε, σε εποχές που γίνονται σπουδαίες αλλαγές ε, στην Ευρώπη, ε, το 2015 είχαμε την πρώτη, τα πρώτα ε, στοιχεία για το κλίμα. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη που προτάθηκα ως Επίτροπος Ενέργειας. Η συνεργασία μου δε μαζί σας, τους Ευρωβουλευτές, θα με επιτρέψει να επιτύχω τους στόχους που έχουμε θέσει όλοι ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Well, Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σίμψον. Ευχαριστώ και σας, συνάδελφοι, για τη συμμετοχή σας. Λίγη εδώ η ακρόαση. Σας θυμίζω ότι θα συνεδριάσουμε ε, με τους συντονιστές το απόγευμα και κλεισμένων των θυρών για να αξιολογήσουμε την παρούσα ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι.